Uh, dear friends, ladies and Φίλοι, κυρίες και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος, με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι έχετε προσέλθει για αυτή τη διήμερη συνεδρία της Επιτροπής μας με διάφορα θέματα. Πριν αρχίσουμε όμως πριν κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης, να δώσουμε το λόγο στους διερμηνείς μας. Πρώτα πρώτα θα πω στα πολωνικά λίγα πράγματα. Όπως γνωρίζετε, το έργο μας ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό θα έλεγα, εξαρτάται από την συνεργασία μας με τους διερμηνείς και τη δράση των διερμηνέων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η πολυγλωσία είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μα και οι διερμηνεί βρίσκονται στην καρδιά των εργασιών μα. Χωρί αυτού δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Και έχουμε μάλιστα το μεγαλύτερο αριθμό γλωσσών παγκοσμίω που μεταφράζονται ταυτόχρονα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν συγκρίνεται ούτε καν με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμεί έχουμε 24 γλώσσε που μεταφράζονται συνέχεια ε, συνεχώς, ίσως όχι σε όλες μας τις συνεδριάσεις, ίσως όχι σε όλες τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σίγουρα στις στην Ολομέλεια έχουμε συνεχώς διερμηνία από και προς 24 γλώσσες. Και οι διερμηνείς είναι οι συνεργάτες μας και θέλουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ τους. Την πιο αγαστή. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους διερμηνείς που θα μας πούν λίγα λόγια κατά την έναρξη της συνεδρίας. Οπότε σας θέρμα παρακαλώ, βάλτε τα ακουστικά σας, γιατί ο καθένας μπορεί στη μητρική του γλώσσα να ακούσει το μήνυμα των διερμηνέων. Γιατί έτσι είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε το λόγο στους διερμηνείς. Η διερμηνή σα πληροφορούν τα λύπης ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία, που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα τη διερμηνίας για του ευρωβουλευτέ και του Ευρωπαίου πολίτε κινδυνεύει. Δυστυχώ, λόγω τη εργασιακή διαμάχη, η διερμηνία θα σταματήσει στις 6.30 ακριβώ, όπως προβλέπει το πρόγραμμα της συνεδρίασης. Okay. Ε, ε, Οπότε σήμερα, λέει ο Πρόεδρος, στις 6.30 δεν θα έχουμε υπέρβαση ωραρίου, γιατί συνήθως παρακαλούμε τους διερμηνείς να παραμείνουν 10-15 λεπτά. Σήμερα δεν ε, είναι εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6.30 ακριβώς. Μερικές φορές ο χρόνος πρέπει να τηρείται. Οπότε, ε, στη, στους τριμερείς διαλόγους έχουμε τεράστιες υπερβάσεις. Ε, ε χρειάζεται μια, μια φορά σε ένα τριμερή διάλογο να κάνουμε υπέρβαση ωραρίου κατά πέντε ώρες. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, ειδικά στους τριμερείς διαλόγους. Ε, και πολλές ε, φορές έχουμε υπερβάσει ωραρίων, όχι μόνο στους τριμερείς ε, διαλόγους, αλλά και στις συνεδριάσεις επιτροπής. Αυτή τη φορά όμως θα τηρήσουμε πολύ πιστά το πρόγραμμα και θα ολοκληρώσουμε στις 6.30 ακριβώς. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη και αν δεν υπάρχουν σχόλια να εγκρίνουμε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν παρακαλώ σχόλια. Όχι. Σημείο 2 Ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσει. Ε, σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 23η και 24η Απριλίου 2018. Αν μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση δεν υποβληθούν παρατηρήσει ή ενστάσει, θα θεωρηθούν ω εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό σημείο τη ημερήσια διάταξη που είναι το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη και που έχει θέμα την ανάπτυξη υποδομών για τα αναλλακτικά κάψιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώρα για δράση. Ο εισηγητής μα είναι ο κύριο Κρασνοντέμσκι, που όπω ξέρετε έχει εκπονήσει γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών, που είναι η αρμόδια κατ' ουσίαν Επιτροπή για το σημαντικό αυτό θέμα τη ανάπτυξη υποδομών για τα αναλλακτικά κάψιμα στην Ευρώπη και σήμερα το απόγευμα. Ο κύριο Τσέσακ, επίση από το ECR, από του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ, αντικαθιστά τον κύριο Κρασνοντέμσκι, που είναι ο εισηγητή μα. Παρακαλώ. Κύριε Τσέσακ, εκπροσωπείτε σήμερα από ό,τι κατάλαβα τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντέμσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ο καθηγητής ο κύριος Κρασνοντέμσκι, δυστυχώς κολλείεται σήμερα γιατί είχε κάποια προβλήματα στη, στην πτήση του και στις ανταποκρίσεις, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει εγκαίρος. Αγαπητοί φίλοι, λέει ο κύριος Κρασοντεύσκη, νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα τη γνωμοδότησή μου για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης ε, και ε, έκανε μια αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων πολιτικής των κρατών μελών, είναι η ώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ε, τονίζοντας τη δική του δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών για τα αναλλακτικά καύσιμα. Δεν θα πρέπει βέβαια να υποτιμούμε άλλες ανταγωνιστικές αγορές, όπως είναι η αγορά της Κίνας για παράδειγμα, που αναπτύσσουν τα δίκτυά τους με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι θα περιμέναμε ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επιταχύνουμε το ρυθμό ανάπτυξης και της δικής μας αγοράς. Γιατί οι δεμοί θα χάσουμε την όθηση και τις δεξιότητες ε, και θα υστερούμε σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Γι' αυτό και εκπώνησα την παρούσα γνωμοδότηση που επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες που αφορούν το ζήτημα των εναλλακτικών καυσίμων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η φωνή της ε, Επιτροπής Ήτρε να εισακουστεί από την Επιτροπή Μεταφορών. Και θα ήθελα και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών να καταλάβουν τη δική μας λογική. Γι' αυτό και θα επικεντρωθώ στα ζητήματα που ενδιαφέρουν κυρίως την Επιτροπή Ήτρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο κυρίως θέματα. Πρώτο, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη για ηλεκτροκίνηση να μην αποβεί εις βάρο ε, τη ασφάλεια του εφοδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε στην ηλεκτροκίνηση. Αλλά οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να συμβαδίζουν με την επένδυση στα εφή δίκτυα και στην ανάπτυξη σημείων επαναφόρτησης. Επίσης, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην έχουμε αύξηση των τιμών της ε, τις ώρες της εχμής της κατανάλωσης. Επίσης, θα πρέπει ε, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα διαθέσιμα κονδύλια και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνέργειες. Έτσι, θα αναπτύξουμε στο έπακρο το δυναμικό των εναλλακτικών καυσίμων, λαμβάνοντα υπόψη το μηχανισμό ε, συνέδρου στην Ευρώπη, ε, τον ορίζοντα για την Ευρώπη και τα διαρθρωτικά ταμεία, που αναπτύ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ορθολογικό συντονισμός μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων και να αποφύγουμε την κοιλάδα του θανάτου που μερικές φορές συμβαίνει μεταξύ την επιστημονική έρευνα την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιτόπου εφαρμογή. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή που δείξατε και περιμένω τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες σας. Όσον ούπο θα υποβάλω και νέες προτάσεις αφού εξετάσω τις τροπολογίες σας και συμβιβαστικές τροπολογίες επίσης. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσέσακ για την ανάγνωση της ε, παρουσίασης του συναδέλφου μας, του καθηγητού του κ. Κρασνοντέμσκι, που είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στους ε, ηγητές. Η κυρία Χένα Βερκούνερ επισκολίεται. κολλείεται. Έστειλε όμως στη γραμματεία της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας τα σχόλιά της, τα οποία θα σας διαβάσω. Madam Henna Virkunen, Shadow Reporter of uh, behalf of EPP uh, Political Group. I would like to thank... Και όδες για το Ευρωπαϊκό Λόγο Κομ να σας ευχαριστήσω κύριε Κραστοντέμσκι για το σχέδιο κειμένου και συμφωνώ με την άποψή σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναβαθμίσουμε τη βιομηχανία μας για να έχουμε τέτοιες ε, μπαταρίες ε, στην ε, Ευρώπη και να υπάρχει τέτοια λυσίδα αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα γιατί είναι πολύ σημαντική η αυτοκινητοβιομηχανία μας. Οπότε έτσι θέλουμε να προαγάγουμε τα αναλλακτικά καύσιμα για τις μεταφορές, να υπάρχει λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και να υπάρχουν λιγότερες ε, ε, ε, επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Θέλουμε να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, οπότε θα πρέπει η Ένωση να τάξει κάποιους στόχους και να υπάρχει τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Θα πρέπει να μετέλθουμε πάνω μέσω για να περιορίσουμε τις εκπομπές και τα αναλυτικά καύσουμε ένας αποτελεσματικός αλλά και γρήγορος ε, τρόπος τόσο ώστε να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές. Οπότε θεωρώ ότι τα βιώσιμη βιοκαύσιμα είναι σημαντική απάντηση όσον αφορά το πώς θα περιορίσουμε τις ε, εκπομπές ε, από τα αυτοκίνητα. Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε επιτυχίες στο μέτωπο της αναζήτησης εναλλακτικών καυσίμων για κάθε είδους μεταφορών και ε, η αγορά ε, δεν έχει αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει πάντως οι λύσεις μας ε, να βασίζονται στην συμπεριφορά της αγοράς. Έχουμε διαφορετικά καύσιμα και χρειάζεται επίσης τα σημεία φόρτισης να είναι προσβάσιμα στο κοινό και θα πρέπει επίσης να ενεργήσουμε για αυτά τα σημεία φόρτιση σύμφωνα με συνθήκε τη αγορα. Άρα χρειάζεται να αναζητηθούν τέτοια ενεργειακά καύσιμα, ούτως ώστε αυτή η τάση να συνεχιστεί με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά ε, μέσα όπως ε, το μέσον ε, Connecting Europe Facility, το Horizon, το SEF. άρα και αυτά αποτελούν τις παρατηρήσεις της ε, κυρίας Βίρκον που είναι ισχυώδης εισηγητρία του ΕΛΚ. Τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες, η κυρία Φέρνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το σχέδιο κειμένου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του δικτύου των εναλλακτικών καυσίμων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Να εντοπίσουμε το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος κλπ. Γιατί χρειάζεται να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Θα πρέπει να έχουμε λύσεις τεχνολογικά ουδέτερες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, έχουμε κάποια εθνικά προγράμματα πλαίσιο τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε γιατί δεν ανταγωνούνται στους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον. Και επίση δεν έχουν επιδείξει όλα τα κατημέλη τόσο μεγάλη φιλοδοξία. Άρα θα πρέπει αυτά να τα αναφέρουμε στην ε, έκθεση. Και αν δεν επαρκούν αυτά τα προγράμματα δράσης, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί προς κάποιο είδους νομοθεσία που να προβλέπει κάποια ελάχιστα δεσμευτικά για τα κράτη-μέλη. Για 12 έως 22 εκατομμύρια μιλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανάγκη επενδύσεων μέχρι το 2022. Για να βρούμε τα χρήματα αυτά από τον ιδιωτικό τομέα δεν αρκεί να περιμένουμε την καλή μας τύχη, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες. Και ακόμα δεν αρκεί. Εμείς προτείνουμε ένα mobility fund το οποίο θα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες μέλη και τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις στους τομείς εκείνους που έχουν προτεραιότητα. Στο ταμείο αυτό μπορεί, μάλλον με το ταμείο αυτό, μπορεί να ε, περιοριστεί κάπως ο επενδυτικός κίνδυνος. Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει ακόμα τη σχετική υποδομή. Και οι υποδομή, αν αυτοί που κατασκευάζουν υποδομές, αναμένουν τους κατασκευαστές. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε, διότι και σε άλλους τομείς διεξάγονται συζητήσεις. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τις κοινότητες και τις κοινοτικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιχειρηματολογήσουν πιστικά ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις στους τόπους όπου βρίσκονται και λειτουργούν. Εάν αναμένουμε μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, τότε σε περιοχές τη υπαίθρου δεν πρόκειται να γίνει απολύτω καμιά επένδυση. Μόνο εκεί όπου υπάρχει ελκυστικότητα για τέτοιες επενδύσει και αυτά είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Εγώ είμαι ωστόσο υπέρ του να λάβουν, του να έχουν την ευκαιρία αυτή και οι επιχειρήσεις που δρώνουν σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου για τα σχόλιά σας. Ο κύριος είναι των ε, Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για να επιτύχουμε τους στόχους του, της Συμφωνίας του Παρισιού πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων στις μεταφορές που είναι και ο μόνο οικονομικό τομέα της Ένωση, όπου από το 1990 έχουν αυξηθεί οι εκπομπέ αυτές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Πάλι η έκθεση παραπέμπει σε στατιστικές που λένε ότι 94% των μεταφορών στην Ένωση εξαρτάται από το πετρέλαιο το οποίο κατά 90% εισάγεται. Τεράστια πρόκληση λοιπόν αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους του Παρισιού και να μειώσουμε τις εκπομπές καυσαερίων στον τομέα των μεταφορών. Πολλοί τρόποι υπάρχουν για να προσεγγίσει κανείς ε, τον στόχο αυτό και χρειάζεται βέβαια ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών. Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας στα αυτοκίνητα, στις δημόσιες μεταφορές, να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάρει το ποδήλατο να πάει στη δουλειά του και βεβαίως συστήματα αποθήκευσης και αποδοτική χρήση της ενέργειας. Όλα αυτά είναι σημαντικές πρωτοβουλίες. Και εν τέλει χρειάζεται περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν επίσης πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ρωμαλαία συστήματα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και βέβαια να βελτιωθεί η χρήση των εφισταμένων υποδομών και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό όμως σημαίνει άφθονο ηλεκτρικό ρεύμα και κυρίως ελεύθερη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς περιορισμούς και τα... να μην υπάρχουν τεχνικά κολλήματα εντός της Ένωσης στην ε, παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το χρειαζόμαστε αν θέλουμε να ενσωματώσουμε περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα στις μεταφορές. Πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε τις τιμές επιτρέποντας περισσότερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να ηλεκτροκινηθεί περισσότερο η κοινωνία μέσω των μεταφορών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδιώξουμε και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την περαιτέρω πορεία της εκθέσεως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντέμψκι, για τη του, για το σχέδιο γνωμοδότησης που επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά σημεία. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο τομέας των μεταφορών είναι αυτός που συμβάλλει κατά κανόνα στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και αναγνωρίζουμε για μια ακόμη φορά ότι αυξάνονται οι εκπομπές από τις, μεταφορέ, μεταφο μεταφορές. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό να φέρουμε τις μεταφορές στο επίκεντρο του αγώνα μας περιορισμού των κλιματικών αλλαγών προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις δεσμεύσεις μας από τη Συμφωνία των Παρισίων. Δηλαδή θα πρέπει να απαλλάξουμε τον τομέα των μεταφορών από τις εκπομπέ διοξιδίου του Αφρικά το συντομότερο δυνατό για να τηρήσουμε τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει διεθνώ. Και σίγουρα τα εναλλακτικά καύσιμα διδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο. Ε, γιατί με βάση το τριμερή διάλογο που ολοκληρώσαμε, ελπίζω, την προηγούμενη εβδομάδα, το 14% των ε, εναλλακτικών καυσίμων ζητάμε μέχρι το 2030. Αν ισχύει αυτό και αν όντω ε, είναι βιώσιμη αυτή, αυτό το στοιχείο, ε, θα πρέπει πραγματικά αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα να είναι φιλοπεριβαλλοντικά, οικολογικά και πραγματικά βιώσιμα. Γιατί αν μιλούμε για εναλλακτικά καύσιμα, δεν μπορεί να ε, ε, παράγονται με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό δεν είναι λύση. Μιλούμε για αναλλακτικά καύσιμα που θα προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, τα αγροκαύσιμα που ε, βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση με τις καλλιέργειες ε, για την παραγωγή τροφίμων ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια ανταγωνιστικότητα. Επίσης έχουμε μια πολύ σημαντική πρόκληση ενώπιό μας, γιατί μιλούμε για την κινητικότητα και όταν ε, μιλούμε για κινητικότητα εννοούμε τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να το πούμε καθαρά και εξάστερα και θέλουμε να λειτουργήσει η πρόταση, θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ε, αυτοκινήτων, να μειώσουμε τη ζήτηση για αυτοκίνητα. Και επίση ε, θέλουμε ανανεώσιμες πηγές που θα πηγαίνουν στα, στα λεωφορεία, στα ποδήλατα, στις μαζικές συγκοινωνίε, για να έχουμε πραγματικά ανανεώσιμες, βιώσιμες ε, ε, μεταφορές. Και φυσικά θέλουμε βιώσιμους ισορρευτές και ανακυκλώσιμους ισορρευτές. Κάτι που είναι απαραίτητο για την ηλεκτροκίνηση. Θέλουμε ένα σύστημα πραγματικά με εναλλακτικά καύσιμα και ανανεώσιμο και βιώσιμο και θα συνεργαστούμε στενά με τον κύριο Κρασφροντέμσκι για να ελοπίσουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχλιτσεκ τώρα, εκ μέρου της ΓΚΟΕ. Ο κύριος Κόχλιτσεκ, αντικαθιστά από ό,τι ξέρω τον κύριο Μπενίτο Σιλουάγκα που κανονικά είναι ο σκιώδης ηγητής της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το σημείο αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των τεσσάρων ε, τρόπων μεταφοράς, γιατί δεν ε, είναι όλοι εξίσου ανεπτυγμένοι οι τρόποι μεταφοράς. Ούτε σε όλους τους τρόπους μεταφοράς μπορούμε να ε, απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς τους στόχους που επιδιώκουμε. Επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αφιερώσει, ε, ε σκοπεύει να αφιερώσει 2 με 25 δισεκατομμύρια, τώρα αυτή είναι πολύ ε, γενικός υπολογισμός που αφορά κυρίως τις οδικές μεταφορές αλλά δεν καλύπτει άλλου τρόπου μεταφορά όπω τι θαλάσσιες μεταφορέ. Γιατί πολλά πλοία χρησιμοποιούν ε, πετρέλαιο. ή υγροποιημένο φυσικό, ίσως το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μπορούσε να αποτελέσει ε, ένα λεκτακό καυσίμο και να μας οδηγήσει εξοικονόμηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ τη χρήση αιωλικής ενέργειας για τις θαλάσσιες μεταφορές, για παράδειγμα. Επίσης, τι γίνεται με τις αερομεταφορές. Θα έχουμε ηλεκτρικούς κινητήρες στα αεροπλάνα. Ε, ή έχουμε πολύ ελαφρά αεροσκάφη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας. Επίσης, στους σιδηροδρόμους λέμε ναι στα, στις ηλεκτρικές σιδηροδρομικές μεταφορές, σίγουρα, αλλά 50% του δικτύου ε, δεν μπορεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο να εφαρμόσει αυτή την ανανέωση. Πώς θα αντικαταστήσουμε τους διζελοκινητήρες ε, ε, με κυψέλες καυσίμου ή με κυψέλες υδρογόνου. Δεν έχουν γίνει καν ε, παρκή πειράματα ή έρευνες. Τέτοιες έρευνες έχουν γίνει για τις οδικές μεταφορές, αλλά όχι για τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες και ίσως η ευκολότερη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε καύσιμα που δεν εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Και από αυτήν την άποψη έχουμε καλές υποδομές για το μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο. Έχουμε ήδη αναπτύξει υποδομές για το προπάνιο και το βουτάνιο. Τώρα ως προς την ηλεκτροκίνηση. Και για την ηλεκτροκίνηση χρειαζόμαστε σημαντικές υποδομές, συσσωρευτές για παράδειγμα, ρευματολήπτες και το καθεξής. Ε, αυτό που δεν έχουμε αναπτύξει αρκετά μέχρι στιγμή είναι οι υποδομές για το υδρογόνο. Θα μπορούσαμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τέτοιες υποδομές στο μέλλον, γιατί σε περίπτωση που έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα για παραγωγή υδρογόνου ή να χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο και στις οδικές μεταφορές με τη μορφή κυψέλων υδρογόνου και υδρογόνου. Ε, θεωρώ ότι η γνωμοδότηση του κ. Κρασοντέμσκι είναι πολύ αξιόλογη και όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις που ακούμε ευπρόσδεκτα. ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα τμήμα των γεωργικών εκτάσεων, το μεγαλύτερο τμήμα των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή τροφίμων και όχι για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ίσως ε, τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικός τρόπος παραγωγής. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, ο κύριος Αλεξάνδρου Βαντιούμ από την Γενική Διεύθυνση ΜΟΦ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι ολοκληρώθηκε αυτό το σχέδιο κειμένου. Πολύ ενδιαφέρον από την άποψή μα, γιατί εξετάζει το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με τι προηγούμενε εκθέσει του Κοινοβουλίου. Οπότε το θεωρούμε πολύ θετικό. Επίση, συμφωνούμε Χρειάζεται να επιταχύνει τους ρυθμούς της σε αυτό το μέτωπο η βιομηχανία. Έτσι μόνο θα φτάσουμε να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες του Γιούγκερ, ούτως ώστε να γίνει πρωταγωνιστής ε, όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, ε, την ψηφική τεχνολογία, η βιομηχανία μας, άρα ο μετασχηματισμός να γίνει πιο γρήγορα. Επίσης να κινητοποιήσουμε πόρους ε, στα πλαίσια του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου και με τα DSO να εξασφαλίσουμε θα είναι πιο ευφύ τα δίκτυα και οι μετρητές θα είναι ευφιέστεροι ούτως υπήρ. Και επίσης χρειάζεται ας θυμηθούμε το να συμφωνηθεί το πακέτο για την καθαρή ενέργεια σύντομα και έτσι να οδηγηθούμε σε αυτούς τους ευφύς μετρητές. Επίσης χρειάζεται ανοιχτή πρόσβαση όσον αφορά την επαναφόρτιση και τα σχετικά δίκτυα. Έτσι θα βοηθηθεί η ηλεκτρονική, η εναλλακτική τέλος πάντων κινητικότητα στην Ευρώπη. Ε, συμφωνούμε επίσης με το πώς το συνδέσατε τα θέματα με τις μεταφορές, με την προτυποποίηση που αναφέρατε. Και εμείς αυτά τώρα τα μελετούμε και ξέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις και τα προβλήματα. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε για τις μεταφορές μαζί με τους οργανισμούς τυποποίησης. Βεβαίως, θα αξιολογήσουμε την οδηγία του χρόνου και επομένω θα δούμε την οδηγία αυτή υπό το φω αυτών των νέων προκλήσεων. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, που μας εξήγησατε την άποψη τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον κύριο Τσέσακ. Αν εκ μέρους του συντάκτη της γνωμοδότησης θα ήθελα να πει δύο λόγια για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για όλες τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν παρουσιάζοντας τις θέσεις των πολιτικών ομάδων και, και ο συνεργάτης μας και εγώ προσωπικά σημειώσαμε με μεγάλη προσοχή όλες τις παρατηρήσεις και τις θα τις διαβιβάσουμε στον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντέμσκι. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ε, η υποβολή των τροπολογιών μπορεί να γίνει μέχρι αύριο 19 του μηνό, μέχρι τις 6 το απόγευμα. 19 έκτου, 6 το απόγευμα. Λίγη διορία για την υποβολή τροπολογιών. Η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2018 ενώ η ψηφοφορία στην αρμόδια κατουσίαν επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Μεταφορών, θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Νοέμβριο. Οπότε μην ξεχνάτε ότι διορία για την υποβολή τροπολογιών έχετε μόνο μέχρι τις 19 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι αύριο 6 το απόγευμα το βράδυ. Σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 5 το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Περιφερειακής, ε, ανα, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σύνοχης, ε, αγροτικής ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο και περικαθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο Συνοχή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού σε ό,τι αφορά στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Η συγκέντριά μας είναι η κυρία Σοφία Σακοράφα από την ΚΟΕ. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης ε, που αφορά την κατάργηση του κανονισμού ε, που τροποποιεί πολλά ε, ταμεία στα πλαίσια του επόμενο πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, υποβάλει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που εγκρίνουν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δηλαδή και υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι ο πρωταρχικό στόχο του συγκεκριμένου κανονισμού. Η πρόταση ε, για την συζήτηση έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοκιμαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεταρρύθμισης και ο μηχανισμός ε, υλοποίηση αποτελεσμάτων για μια πιλωτική περίοδο ε, πειραματική, δηλαδή για τα διετία 2018-2020. Για όσοι ενδιαφέρονται, αύριο η αρμόδια κατουσία Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα οργανώσει αύριο ακρόαση για το θέμα αυτό. Αύριο δηλαδή η Επιτροπή Ρέγγι θα διοργανώσει σχετική ακρόαση. Όσοι πιστοί προσέλθετε και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν να δώσω το παρόν αύριο στην σχετική ακρόαση της Επιτροπής Ρέγγι. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, στην κυρία Σακοράφα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διάψευσης των επικρίσεων και ενίσχυσης της αιτιολόγησης και της λογοδοσίας των δαπανών των Ταμείων Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετήθηκε στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ένας ενισχυμένος προσανατολισμός της επιδόσεις. Συγκεκριμένα για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίστηκε ένα πλαίσιο επιδόσεων όπου περιγράφονται λεπτομερώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τι επενδύσει και ο τρόπο μέτρηση προόδου που σημειώνεται στην πορεία προ την επίτευξη των ε, στόχων που έχουν μπει. Μέχρι το 2019 θα διενεργηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων και τα προγράμματα που θα έχουν επιτύχει τα ορόσημα και του στόχου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο αποθεματικό επίδοση που, όπω ξέρετε, πρόκειται για το 6% των πόρων που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, ενώ όσα θα έχουν αποτύχει ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την επιβολή κυρώσεων. Η συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής τροποποίησης με εξέπληξε προσωπικά δυσάρεστα. Εν ολίγης, καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν εθελοντικά, εν όλο ή εν μέρη, τη διαχείριση των πόρων του αποθυματικού επίδοση στην Επιτροπή, προκειμένου να στηρίξει όπως διακαώς επιθυμεί οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κατά την προσωπική μου άποψη, η πολιτική συνοχή και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν μοιράζονται και δεν εξυπηρετούν του ίδιου στόχου. Οι εκ των προτέρων καθώ και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα συνιστούν μείζωνα κίνδυνο για την επίτευξη τη βιώσιμη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η σύνδεση τη πολιτική συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την επίτευξη των στόχων τη όπω ορίζονται στι συνθήκε. Για τον λόγο αυτό, η μετατόπιση επιπλέον 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι το συνολικό αριθμητικό μέγεθο για το αποθεματικό επίδοση, για την εξυπηρέτηση στόχων που συνδέονται στενά με την διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, αποτελεί σαφή παρέκκληση από τον κύριο σκοπό της πολιτικής για τη συνοχή, δηλαδή την μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Ο επαναπροσανατολισμό ενό τόσο σημαντικού μέρου των πόρων θα διαταράξει την εφαρμογή και θα επηρεάσει αρνητικά τον αντίκτυπο τη πολιτική συνοχή κύριες και συμπληρωματικές αρχές της, όπως η αλληλεγγύη στην πράξη, η εύλογη και δίκαιη ανακατανομή του πλούτου, καθώς και η ίδια λογική που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για την επίτευξη επιδόσεων, θα υπονομευθούν σοβαρά. Όσον αφορά το διαδικαστικό σκέλος, θεωρώ ότι η πρόταση έρχεται με καθυστέρηση και είναι εξαιρετικά ασαφής η σχετική τροποποίηση θα έχει αναδρομική ισχύ, ενδεχομένως θα προκαλέσει δημοσιονομικές διαταραχές επί των συμφωνημένων εθνικών αιτήσεων δόσεων και είναι πιθανό να θέσει έναν αμφιβόλο ήδη προγραμματισμένες δαπάνες για συγκεκριμένα έργα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν και είμαι υπέρμαχο των μεταρρυθμίσεων, θα αποδοκιμάσω για μια ακόμη φορά του χρηματοδοτικού μηχανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει με αποκλειστικό επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την οικονομική διακυβέρνηση κατά τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Όπω γνωρίζετε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ανακατανομή των κονδυλίων τη συνοχή προ όφελο του προγράμματο στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ η Επιτροπή προτείνει τώρα μια εκ νέου σημαντική αύξηση τη συνολική τη χρηματοδότηση φαίνεται ότι το χρηματοδοτικό ισοζύγιο ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και την οικονομική διακυβέρνηση θα επιδεινωθεί κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο. Η Επιτροπή προτείνει μεν τη θέσπιση ενό νέου προγράμματο στήριξη των μεταρρυθμίσεων περίπου ύψου 21 δισεκατομμύριων ευρώ, με χρηματοδότηση από το μέσο ευελιξία και σε πλήρη διαχωρισμό από τα ευρωπαϊκά διαθροτικά και επενδυτικά ταμεία. Εν τούτης, παράλληλα, σχεδιάζει σημαντική μείωση της συνολικής χρηματοδότησης για τη συνοχή. Κλείνοντα λοιπόν την αρχική μου τοποθέτηση, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ενώ η επιμερισμένη διαχείριση που αποτελεί τον κανόνα για τη διαχείριση των πόρων τη συνοχή δημιουργεί την εντύπωση μια συνδιοκτησία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απόφαση ενό κράτου μέλου να χρησιμοποιήσει εν μέρη ή στο σύνολο το αποθυματικό επίδοση για την υποστήριξη των διαστατικών μεταρρυθμίσεων σηματοδοτεί, όπω σαφώ προτείνεται, τη μετάβαση σε καθεστούς άμεσης διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα χάσουν τον έλεγχο επί των σχετικών πόρων, ενώ κάθε πρόταση για την ανάληψη μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων θα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα αξιολόγησης, έγκρισης και διαχείρισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να καλέσει την Επιτροπή Ρέντζη, αρμόδια επί και τις Επιτροπές ΕΚΟΝ και ΜΠΑΝΤΣ ως συνδεδεμένες επιτροπές να απορρίψουν την πρόταση της Επιτροπής. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, madam. Σας ευχαριστούμε κυρία Σοκοράφα. Ακούσαμε τις παρατηρήσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης. Θα περάσουμε τώρα στους γεώδεις ηγητές. Ο κύριος Κρίστιαν Σίλβιο Μπουσόη, που είναι ο σκιώδης ηγετής του ΕΛΚ, κανονικά έπρεπε να λάβει το λόγο, αλλά απουσιάζει και μου ζήτησε να διαβάσω τις παρατηρήσεις του. Τι γράφει λοιπόν ο Κρίστιαν Μπουσόη. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το μέλλον της πολιτικής αυτής, της πολιτικής συνοχής και, της αρχή, και την αρχή της συζήτησης για ε, την Ευρώπη με, τα, με το νέο πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο και εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις ε, του προγράμματος ε, στήριξης ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Οι εθνικές μεταρρυθμίσεις της κεφαλαγορές και στην αγορά εργασίας, στη δημόσια διοίκηση, στη φορολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητες στα κράτη-μέλη το νέο πρόγραμμα στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων θα διαδραματίσει νευραλγικό ρόλο στην μελλοντική εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμίσεων. Και χαιρετίζω τις ε, διατάξεις που θεσπίζονται στο ΠΔΠ μετά το 2020. Δηλαδή, κάθε ε, εργαλείο θα πρέπει να έχει το ξεχωριστό δημοσιονομικό κονδύλιο από, το, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Από την άλλη πλευρά, το ευρωπαϊκό, τα, προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα της πολιτικής συνοχής έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής την πιο ορατή προστιθέμενη αξία. Και εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών, η πρόταση ανακατεύθυνση σημαντικού αριθμού κονδυλίων από το Ταμείο αυτό και από την πολιτική συνοχή θα επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο την απήχηση της πολιτικής, αλλά και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα της πολιτικής. Και ως εκ τούτου μπορούν ε, να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ευρωσκεπτικιστική θέση, αν ε, περικόψουμε ακόμη περισσότερο την πολιτική συνοχής μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Ρέγγι, ε, στηρίζω την έκκληση της κυρίας ε, Σακοράφα να απορρίψουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά μας λέει ο σκιώδης ηγετής του ΕΛΚΟ, κύριος Κρίσιαν Σόι. Ακούμε τώρα το σκιώδη εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον κύριο Γιένς Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό ότι διαμορφώνεται συνένεση στην Επιτροπή μας, διότι η σύσταση που θα κάνω στην πολιτική μου ομάδα προς την ίδια κατεύθυνση κατευθύνεται, δηλαδή να αποδεχθούμε την πρόταση της κυρίας εισηγήτριας. Τους λόγους τους εξήγησε και η υπόδειξη του χριστιανοδημοκράτη συναδέλφου μας ότι θα πρέπει να διατεθούν ήδη οι πόροι και αυτό το βρίσκω σωστό. Δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση όταν οι πόροι της Ένωσης στηρίζουν με τον σωστό τρόπο, το τονίζω αυτό, τις προτάσεις του προγράμματος πλαισίου. Αυτά που προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα υποστήριξης να πάνε δηλαδή σε direct management που σημαίνει να μην συνδέονται με τις προσπάθειες των χώρων μελών και τα χρήματα αυτά, να, τα κονδύλια αυτά να αφαιρούνται από το Περιφερειακό Ταμείο, αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό και επομένω λάθο. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμών και στην τελευταία συζήτηση δεχτήκαμε τη δημιουργία του αποθεματικού μονάχα με μεγάλη δυσαρέσκεια διότι στην ουσία πρόκειται για περικοπή. Και τα χρήματα από το αποθεματικό απόδοσης ξεφεύγουν από τις χώρες μέλη που έχουν ωστόσο καταβάλει προσπάθειες. Δηλαδή έρχεται αντίθετη πλέον εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς που δεν μπορώ να δεχτώ. Στα πλαίσια του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Και εκεί όμως ισχύει ότι η στάση της δικής μου πολιτικής ομάδας θα είναι ότι θα πρέπει να σημούν αυτά με πρόσθετα κονδύλια. Και το τελευταίο επιχείρημα που κατά τη γνώμη μου δεν έχει τεθεί ακόμη είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πολύ λίγο χρόνο πλέον στα πλαίσια του παρόντος ΠΔΠ για να προωθήσει τις προτάσεις αυτές. Και είτε πρέπει να το κάνει στη βάση αξιολόγηση που έχει ήδη γίνει και όπου οι χώρε μέλη δεν έχουν πλέον καμία δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτήν, είτε για αυτήν που θα γίνει ακόμη, δηλαδή τέλη του 2019, που σημαίνει ότι θα είμαστε πλέον μόνο 12 μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου πολίτου δημοσιογραφικού πλαισίου. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή την προσπάθεια. Μου φαίνεται δηλαδή λίγο σαν μια τέτοια, τέτοιες σημαντικές αλλαγές να γίνονται με σαλαμοποίηση, δηλαδή φέτα-φέτα. Και δεν συμφωνούμε. Έτσι λοιπόν, στήριξη προς την εισηγήτρια για την αναπομπή της πρότασης. Uh, thank σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε. Η κυρία Βιέρινγκ των Φιλελευθέρων. Άλντε. Ήρθατε ακριβώς στη σωστή στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ακριβέστατοι. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα κύριε Πρόεδρε. Είχα άλλε υποχρεώσεις στο Κοινοβουλίο. Σα ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσά, κυρία Σακοράφα για το σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με τι αρχέ τη προτάσεω τη Κομισιόν. Μέσα στην ΑΛΔΕ εμεί καταρχήν συμφωνούμε με την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πιο ευέλικτο τρόπο. Έτσι λοιπόν καταρχήν είμαι υπέρ τη προτάσεως τη Κομισιόν. Βέβαια υπάρχει και ένα αλλά. Έχω κάποιε ερωτήσει ακόμα σε ό,τι αφορά τον χρονισμό, το timing την εκτέλεση των διαφόρων δαπανών και την αιρεσιμότητα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευκρινιστεί μέσα στην πρόταση με ορισμένε τροπολογίε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τα εξή. Τι κόστο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ε, αποθεματικό απόδοση. και σε σχέση με αυτό πώ θα διασφαλίσετε ώστε οι χώρε μέλη να μπορέσουν να λάβουν τα έξτρα κονδύλια, θα έχει χρήματα. Εννοώ δηλαδή. Σε τι θα πρέπει να στοχεύσουμε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο πώς αντέδρασαν οι χώρες μέλη στις απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις αλλαγές, για τις μεταρρυθμίσεις. Ό,τι αφορά το χρονισμό της προτάσεως, διαρωτώ με ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πώς θα εκτελεστεί το νέο αυτό project και πώς το βλέπουμε σε συσχετισμό με, το, με τις προτάσεις για το επόμενο πι. Ελπίζω να μπορέσουν να συζητηθούν αυτές οι ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπήρχαν και άλλες προτάσει από όλε τι πολιτικέ ομάδε, πολύ ευρύτερε από αυτές που είπατε εσείς. Τώρα πάντως έχετε η ώρα για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναλάβει να το πράξει ο κύριος Μιγγέλ Χιλτέρχε από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε, Πρόεδρε. Η αφετηρία για αυτή την πρόταση είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις... Συγγνώμη, με ακούτε τώρα καλύτερα? Α, μάλιστα. Έλεγα ότι η βάση για την πρότασή μα, η αφετηρία τη είναι ότι αυτέ οι διαδοτικέ μεταρρυθμίσει είναι μια προπόθεση για την ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να προβούμε σε επενδύσει, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε πλήρη αποτελεσματικότητα ε, και το να πιάσει τόπο τέλο πάντων η επένδυση εάν ε, δεν υπάρχει η σωστή ε, νομοθεσία και δεν είναι αποτελεσματική η διοίκηση. Οι ευρωβουλευτές έχουν καταλάβει ότι υπάρχει αυτή η πιλωτική φάση στα πλαίσια του πολιτούς τωρινού πλαισίου και για το επόμενο πολιετές πλαίσιο έχουμε προβλέψει διαφορετικές προϋποθέσεις και ρυθμίσεις. Να σας πω για την πιλωτική φάση τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περικοπή όσον αφορά τα κονδύλια. Αυτό είναι το σημαντικό μας μήνυμα. Και για τον κανονισμό CPR έχουμε επιφέρει κάποιες τροποποίησεις. Δηλαδή μπορεί να ε, επιστρατεύσει αυτό το απόθεμα των επιδόσεων για να υποστηριχτούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει αυτό το επαθεματικό. Εάν τα κράτη-μέλη θέλουν να τα πράγμα να μείνουν όσοι έχουν μπορούν να αναλώσουν αυτό το αποθεματικό σε συγκεκριμένα έργα ή προγράμματα. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό σε αυτή την πιλωτική φάση και είναι σημαντικό το ότι δεν υπάρχει κάποια αντίθεση, σύγκρουση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο πρέπει να υπάρχει συνέπεια και εμείς έτσι στηρίζουμε τις επενδύσεις. Οπότε και έτσι θέλουμε να διαμορφωθεί το μελλοντικό μοντέλο της ανάπτυξης. Δεν προτείναμε εμείς τις μεταρρυθμίσεις. Τις προτείνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι εύστοχες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, να αφορούν κάποια προβλήματα που έχουν επισημανθεί κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, άρα θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με την Κομισιόν για να μπορούμε να επισημάνουμε ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι τους και έτσι να αξιοποιηθεί αυτή η πιλωτική φάση με το να δράσουμε ταχαίως. Περί του θέρος θα ξέρουμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη με το αποθεματικό και για αυτή την προγραμματική περίοδο θα ξέρουμε τι θα ισχύσει. Αυτή είναι η πιλωτική φάση. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε υποβάλει την πρότασή μας για έναν κανονισμό ε, που θα αφορά αυτό το πρόγραμμα υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων. Θα υπάρχει αυτό το εργαλείο επιδόσεων και επίσης βαθμίσουμε την τεχνική αρρωγή και ένα νέο εργαλείο διευκόλυνσης για την σύγκληση όσον αφορά τα κράτη-μέλη που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Τώρα, για το επόμενο πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό το εργαλείο επιδόσεων της μεταρρύθμισης. Εδώ έχουμε ε, από τη μία μεριά 11 δις για τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την κλίδα συνοχής διατίθεται αυτό για αυτές τις μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και όσο κρατημέλη δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους διαθέσιμους πόρους, τότε θα πάνε σε κάποιο είδου ε, κοινό κορβανά, κοινό κουμπαρά, οπότε να αξιοποιηθούν έτσι οι πόροι εν είναι σημαντικό να περάσει αυτό το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάποιο είδου ε, διαφορετική χρήση των πόρων. Εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι οι προποθέσει για το να πιάσουν ε, ε, τόπο οι πόροι των ευρωπαϊκών επενδύσεων θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε δημοσιονομική στήριξη και το κράτος μέλος το οποίο παίρνει αυτή την πρικοδότηση να μπορεί να τα αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα για τις ε, μεταρρυθμίσεις όσον αφορά αυτού του είδους τη διαρθωτική πολιτική. Κύριε Σακοράφα, ω εισηγήτρια της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ, έχετε το λόγο ούτως ώστε να κάνετε τη σύνθεση των παρατηρήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους και τις τυχόν παρατηρήσεις που είχαν και θα μου επιτρέψετε επίσης να απευθυνθώ στην Επιτροπή και να της υπενθυμίσω ότι η συγκεκριμένη πρόταση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση με τις πρόσφατες δηλώσεις Επιτροπής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας υπενθυμίσω ο κύριος Χαν στις 15 Μαρτίου του 2018 απαντώντας σε επερώτηση παρότρινση Επιτροπής Ρέτζη για την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης και κατανομής του αποθεματικού επίδοσης, τοποθετήθηκε αρνητικά, αναφέροντας επιλέξει τα δυνητικά ωφέλη από την προτινόμενη τροποποίηση επίσπευση είναι σημαντικά λιγότερα από τα μειονεκτήματα, όπω ο διοικητικό φόρτο, η πολυπλοκότητα, η έλλειψη συνοχή σε όλα τα κράτη-μέλη και τα προγράμματα και οι μη προγραμματισμένε αλλαγές στην ενδεικτική δημοσιονομική πορεία. Η πρόσθετη εργασία των νομοθετών για τη μιας μια πιθανή τροποποίηση προστίθεται σε αυτό. Αυτά είπε ο κύριο Χάν στην Ολομέλεια. Δεν μπορώ λοιπόν να αντιληφθώ πώς η τροποποίηση περί της επίσπευσης είναι εν καταστροφική και πώς αυτή που προτείνει η ίδια η Επιτροπή για την αλλαγή του προσανατολισμού και του τρόπου διαχείρισης του αποθεματικού επίδοσης είναι απόλυτα θεμητή και επιθυμητή. Πρόκειται λοιπόν για μια σαφή περίπτωση εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών, θα μου επιτρέψετε να πω. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που στην συζήτηση που έγινε οι περισσότερες ομάδες συμφωνούσαμε απόλυτα ε, για την, ε, σε ό,τι αφορά την, τρο, ε, την προτινόμενη τροποποίηση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να καλέσω την Επιτροπή να αποσύρει άμεσα την παρούσα πρόταση, να μας απαλλάξει από την πρόσθετη εργασία της τροποποίησης και να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρώτη εφαρμογή του πλαισίου επιδόσεων. Σας ευχαριστώ. Thank you, madam. Σας ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λίγη αύριο 19 Ιουνίου στις 6. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας Ήτρε θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Και στην αρμόδια καθήλη Επιτροπή τη Ρέγκη και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχουν ακόμη ε, επιβεβαιωθεί με ημερομηνία. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και να καλωσορίσουμε τον κύριο Κάλλος Μοέντας, τον ε, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία. Η ανταλλαγή απόψε μαζί του θα γίνει στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου και θα συμπεριλάβει τα νεοθεσπιθέντα νομοθετικά προγράμματα στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα θέλαμε να συζητήσουμε με τον Επιτροπό αφού ακούσουμε την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon Ευρώπη, Europe, τα ειδικά προγράμματα του Horizon Europe και το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για την περίοδο 2021-2025. Όπως γνωρίζετε, έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις πριν από δύο-τρεις μήνες, περισσότερες στην δική μας Επιτροπή και είχαμε και κάποιες άτυπες συναντήσεις μελών της Επιτροπής Ήτρε με τον Επίτροπο Μοέντας στο Στρασβούργο, κάτι που ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικό και χρήσιμο. Τώρα έχουμε ήδη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτοιμη και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην τελική συζήτηση τελική φάση της συζήτησης πριν εκπονήσουμε τα σχέδια εκθεσής μας και πριν περάσουμε στο πολιτικό έργο και τη συζήτηση του περιεχομένου του προγράμματος ε, Horizon Europe. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, Γέζη Μπούζεκ, αγαπητά μέλη, χαίρομαι πάντα κάθε φορά που έρχομαι στην Επιτροπή Έρευνας και βιομηχανίας. Και μάλιστα ε, μερικές φορές είναι δύσκολο να προετοιμαστώ γιατί έρχομαι τόσο συχνά στην Επιτροπή σας που νομίζω σας τα έχω πει όλα για το πρόγραμμα Horizon Europe. Πριν μάλιστα την ε, έγκρισή του. Έχω την αίσθηση ότι κάλυψα όλα τα σημεία και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι μια και σας ήδη έχω ενημερώσει σε προηγούμενο στάδιο. Αλλά χαίρομαι που θα σας κάνω σήμερα και την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Horizon Europe. Καταρχήν, ε, να δούμε κάπως γενικά τον προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω κάτι που όλοι γνωρίζετε. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα γιατί θα έχουμε πια λιγότερες χώρες που θα συμβάλλουν, αλλά σε περισσότερες προτεραιότητες. Οι λιγότερες χώρες είναι έτοιμες να αυξήσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό και όλο ε, περισσότερες χώρες ζητούν αύξηση των παραδοσιακών πολιτικών. Οπότε οι συνθήκε ήταν ιδιαίτερα αντίξωε και δυσχερεί. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ε, χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Γιατί καταφέραμε να έχουμε ε, το συμβολικό νούμερο, το, το τριψήφιο, 100 δισεκατομμύρια πακέτο. Και μάλιστα το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι από τα λίγα υπάρχοντα προγράμματα που έλαβαν την προτεραιότητα για αύξηση του προπολογισμού. Καθαρά και εξάστερα. Και μπορούμε να εξετάσουμε με διαφορετικό τρόπο ε, τα νούμερα, αν έχουμε την ευρατόμη ή όχι, αν έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα εντός ή εκτός. Πάντως η αύξηση μεσα εντό η εκτος παντως εντυπωσιακή. Και αν δείτε τα 77 δισεκατομμύρια που ήταν αρχικά το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη και αν βγάλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί θα έχουμε πια 27 χώρες, τότε θα είχαμε 67 ε, δισεκατομμύρια. Οπότε από τα 67 δισεκατομμύρια περάσαμε στα 100 δισεκατομμύρια, σχεδόν 50% αύξηση. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την σημαντική αύξηση. Βέβαια θα με ρωτήσετε, αρκεί, εσεί είστε ικανοποιημένο, είστε ευτυχεί. Όχι, φυσικά δεν είναι επαρκή αυτή η αύξηση και πολύ θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και την επιστήμη. Αν όμως με ρωτάτε αν ε, με ικανοποιεί, με χαροποιεί αυτό το ποσό, τα 100 δισεκατομμύρια, σας διαβεβαιώ ότι είμαι υπερήφανος και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το ποσό. Γιατί γνωρίζω ποιο ήταν το σημείο αφετηρίας και πού φτάσαμε. Και χαίρομαι για τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουμε όλοι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ποια πλευρά θα ταχθώ εγώ όταν θα ξεκινήσουν αργότερα οι συζητήσεις ε, στο εξάμεινο. Τώρα, για το προϋπολογισμό τελευταίο σχόλιο. Προτάθηκε η κατανομή ανάλογα με τους πυλώνες. Μερικοί βέβαια θα προτιμούσαν περισσότερα κονδύλια στον πρώτο πυλώνα, άλλοι θα ήταν υπέρμαχοι του δεύτερου πυλώνα, άλλοι θα προτιμούσαν χρήματα περισσότερα στον τρίτο πυλώνα και κατά πάσα πιθανότητα όλοι έχετε δίκιο. Γιατί Σίγουρα θα χρειαζόμασταν περισσότερα κονδύλια σε όλους τους πυλώνες, αλλά καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε κάποιες ε, επιλογές. Και νομίζω ότι οι επιλογές μας ήταν πολύ ισορροπημένες και λογικές και τη χάνουν της ε, υποστήριξης των συναδέλφων επιτρόπων. Και είμαι υπερήφανος για τις επιλογές τελικά που κάναμε. Τώρα, αν ρίξουμε μια ματιά, ε, καταρχήν, στον πρώτο πυλώνα, ανοιχτή επιστήμη. Πρόκειται για ένα πυλώνα που έχει 25,8 δις που θα εξασφαλίσει τη σημαντική συνέχεια του προγράμματος Horizon 2020 και θα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, πολύ σημαντικά, από τα 13, κάτι δισεκατομμύρια, φτάσαμε στα 17 περίπου δισεκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αύξηση και θα μας καθιστά υπερήφανος. Επίσης, οι δράσεις Μαρή ε, Κιουρί ενισχύθηκαν για τις ε, υποδομές της έρευνας. Επίσης, ε, ανταγωνιστικότητα βιομηχανική, 52,7 δισεκατομμύρια. Επίσης, έχουμε τις προκλήσεις της κοινωνίας για τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση από τα πάνω προς τα κάτω και έχουμε έξι άξονες. Ο πρώτος είναι η υγεία, ο δεύτερος ε, κοινωνία χωρίς ε, αποκλεισμού και ασφαλής, το τρίτο είναι ψηφιακός κόσμος και βιομηχανία, μετά κλίμα και ενεργειακή κινητικότητα και πέμπτος άξονας, τρόφιμα και φυσική πόρη. Αυτοί οι τομείς ε, στόχο έχουν μία διατομιακή, διακλαδική προσέγγιση και διασυνοριακή συνεργασία. Κάτι που είναι και ιδιαίτερα προσφυλέ σε μένα. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ προτάσω την ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε καινοτομίε και καινούργια επιτεύγματα μόνο χάρη σε συντονισμό, συνεργασία διατομεακή, διακλαδική και συντονισμό των πολιτικών. Και γι' αυτό καταλήξαμε στην ιδέα των αποστολών. Θα είμαι σαφής σήμερα, γιατί μερικοί με ρώτησαν ε, πώς βλέπω τις αποστολές και πόσες θα είναι. Η ιδέα είναι απλή θα πρέπει σε αυτόν τον προϋπολογισμό του δεύτερου πυλώνα να δούμε τις αποστολές που θα έρχονται από παντού, γιατί ε, δεν ε, αποκλείονται από το δεύτερο πυλώνα. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτές τις αποστολές. Έχουμε 5 με 10 δισεκατομμύρια ε, αυτό που προβλέπουμε για τις αποστολές στο δεύτερο πυλώνα. 5 με 10 δις. Και αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι το εξής. Καταρχήν θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα κριτήρια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κριτήρια νομίζω ότι είναι πολύ καλά διατυπωμένα στην πρόταση. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν συμφωνήσουμε για τα κριτήρια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις αποστολές. Δεύτερον, μετά τη συμφωνία σας για τα κριτήρια, θα πρέπει να εξετάσουμε τους τομείς των αποστολών. Σε ποιους τομείς θέλουμε αυτές τις αποστολές. Στην υγεία, στην ενέργεια, στην καθαρή ενέργεια, στον καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε σαφείς τομείς δράσεων και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτούς τους τομείς. Προηγουμένω όμω θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα κριτήρια πριν περάσουμε στη συζήτηση για του τομεί. Και ήδη είχαμε πολύ αξιόλογέ συζητήσει, πολύ ενδιαφέρουσε με πολλού από εσά. Μιλήσαμε για τον καρκίνο για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη και μιλήσαμε με πολλούς ευρωβουλευτέ που είναι υπέρ μια αποστολή για τον καρκίνο και νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Οπότε μπορούμε από το Σεπτέμβριο να προσδιορίσουμε αυτούς τους πιθανούς τομείς και στις αρχές του 2019 θα πρέπει να τους προσδιορίσουμε. Και έχουμε και τον τρίτο πυλώνα της ανοιχτής καινοτομία. Για πρώτη φορά έχουμε αυτήν την ιδέα της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και νομίζω ότι θα συνεργαστούμε ώστε το τομέα της καινοτομίας και το EIT και ε, μου στείλατε επιστολή για, την, για το EIT γιατί πολύ συχνά με ρωτάτε ποιος είναι ο ρόλος του EIT. Νομίζω ότι ο ρόλος είναι σαφέστατος. Θα είναι σημαντικός φάρος για την κατάρτιση και για τη δημιουργία του οικοσυστήματος. Τώρα, η χρηματοδότηση, η χρηματοοικονομική υποστήριξη δεν είναι από το EIT, από το, e- αλλά από το EIC. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό τμήμα, σημαντικά τμήματα του οικοσυστήματος. Ό,τι αφορά την επιστολή που έστειλε ως απάντηση για αυτούς που με ρώτησαν για το EIT, να πω ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο προπολογισμό του η ΑΕΤ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογία, 3 δισεκατομμύρια και επίση ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας ε, θα είναι εγκάρσιο, θα υποστηρίζει όλου του πυλώνας. πολύ συχνά μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Καινοτομία. Νομίζω ότι η νέα πρόταση είναι πολύ φιλόδοξη και περιλαμβάνει νέα στοιχεία. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία που μέχρι στιγμή ίσω ε, δεν ε, ανέπτυξα γιατί έχω μιλήσει γενικώ για το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο καινοτομία, αλλά όχι ειδικά. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει το ERC, ε, που ξεκινάει από την θεμελιώδη έρευνα μέχρι την εφαρμογή και μετά έχουμε το EIC, που είναι το Pathfinder, ε, που θα μιλάει για την καινοτομία, για τους ε, καινοτόμους ερευνητές και θα είναι και επιταχυντής. Επιταχυντής για καινοτόμες νεοφύης επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε έχουμε το ERC, Bottom Curiosity, Proof of Concept, Pathfinder και Accelerator. Όλο αυτό είναι το φάσμα της καινοτομίας και περνάμε από τις άκαμπτες επιδοτήσεις σε πιο ευέλικτες και άμεσες επιδοτήσεις που μπορεί να διακόπτονται ή να αλλάζουν. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσά για διαφορετικούς λόγους μου ανέφερα την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών και την ΤΑΡΠΑ. Δεν θα πρέπει να αντιγράφουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες να τις μιμούμαστε τυφλά. Απλώς να αντιγράφουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχουν αποφέρει επιδόσεις. Και το θέμα της ΔΑΡΠΑ, ότι είναι ευέλικτη, μπορεί να διακόψει μια επιδότηση και να περάσει από τη μία στην άλλη, είναι πολύ καλή ιδέα. Και άλλη ιδέα του ΔΑΡΠΑ είναι ότι έχουν τους μάνατζερ των προγραμμάτων, τους υπευθύνους προγραμμάτων και έτσι έχουν πολύ ελαστικούς ε, και καλούς εμπειρογνώμονες που έχουν ε, ε, πολύ εμπεριστατωμένες γνώσεις για το τομέα αυτό και μπορούν πραγματικά να ε, είναι σημείο επαφής μεταξύ όλων των καινοτόμων. Οπότε αυτός ο πυλώνας θα διασυνδέεται με τους άλλους και θα συμπληρώνει κάποιες δραστηριότητες για να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ε, η ιδέα μας ήταν να διπλασιάσουμε και μάλιστα προτεργάτη της πρότασης αυτής ήταν ο κύριος Μπούζεκ να έχουμε κοινή χρήση της αριστείας ε, και να επεκτείνουμε και να αξιοποιούμε από κοινού όλα τα, όλους τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχουμε. Και ο, ο πρόεδρος Μπούζεκ ήταν ο πρώτος που πρότεινε αυτόν τον διαπλασιασμό του προϋπολογισμού και επιτέλους το καταφέραμε. μπορείτε να είστε περήφανος κύριε Πρόεδρε. Και αυτό είναι σημαντικό για όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο για αυτές που δέχονται αυτούς τους μηχανισμούς. Επίσης, ε, μια και ο χρόνο τρέχει, δεν θα σταθώ λεπτομεριακά σε όλα τα επιμέρου σημεία, θα τα αφήσω για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Να πω μόνο δύο λόγια για δύο πολύ σημαντικά πράγματα που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Το ένα αφορά τις εταιρικέ σχέσεις. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές εταιρικέ σχέσεις που έχουν διαφορετικές ονομασίες, αλλά σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι απλούστερο. Και πώς θα το καταφέρουμε θα πρέπει καταρχήν να είμαστε ανοιχτοί προς τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ή με ιδρύματα και έχουμε τρία είδη ρυθμίσεων. Έχουμε τα τις εταιρικές σχέσεις ε, των προγραμμάτων, όπου συνεργαζόμαστε αλλά κάθε τέρος ε, έχει τη δική του χρηματοδότηση. Δεύτερον, έχουμε τις συγχρηματοδοτούμενες εταιρικέ σχέσεις, όπου έχουμε κοινή συγχρηματοδότηση για να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα. Και τρίτον, είναι οι θεσμικές εταιρικέ σχέσεις, όπως το πρίμα και άλλες γνωστές θεσμικές εταιρικέ σχέσεις, τα άρθρα 185 και 187 για παράδειγμα. Οπότε έχουμε μια πλούστευση των εταιρικών σχέσεων. Και ελπίζω να μπορέσουμε αργότερα να περάσουμε σε πιο διεξοδική συζήτηση. Και τέλος, συνέργειες. Πριν ε, ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σας πω ότι κάναμε κάτι πραγματικά ρηξικέλευθο για τις συνέργειες. Σε ό,τι φορά τη σφραγίδα αριστείας, ε, θα περιχαρακώνει και το Horizon Europe και την νομοθεσία για τα διαρθρωτικά ε, ταμεία. Οποιοδήποτε σχέδιο έχει δυνάμει του ορίζοντα Ευρώπη τη φραγίδα αριστεία θα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Με όχι πλέον αξιολόγηση, με του ίδιου χρηματοδοτικού ε, συντελεστέ και εξαιρούνται από τους, νόμους, από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και μάλιστα συμφωνεί ο Επιτρόπος Ανταγωνισμού γι' αυτό. Επίσης, μπορούμε να έχουμε συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε τα Aeronets που έχουν 30% ε, χρηματοδότηση από το ορίζοντας 2020 και 70% εθνική χρηματοδότηση. Τώρα θα μπορείτε να συνδυάζετε τα κονδύλια του ορίζοντας Ευρώπη με τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Κάτι που στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα γίνεται πολύ πιο εύκολο. Οπότε, πρόεδρε Μπούζεκ, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα έχω την ευκαιρία στη συζήτηση να αναπτύξω πιο διεξοδικά κάποια σημεία. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που με καλέσετε. Έχουμε και το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Πακέ. και σας διαβεβαιώ ότι και η Γενική Διεύθυνση και το δικό μου γραφείο είναι στην απόλυτη διάθεσή σας για συζήτηση ε, γιατί πραγματικά αυτή είναι δύσκολη και για όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, μέσω του Γενικού Διευθυντού όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, με καθιστά ιδιαίτερα ικανοποιημένο και χαρούμενο και είμαι στη διάθεση για την περαιτέρω συζήτηση. Εμεί ευχαριστούμε για την προσφέση επιτροπή. Έχετε δίκιο. Τα έχουμε πει επανειλημμένα. Έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά το ίδιο θέμα. Αλλά ακόμα βρίσκεται τις τραπέζες. Ε, όμως η συζήτηση δεν είναι η ίδια γιατί πρόκειται για ένα ζωντανό πρόγραμμα το οποίο συζητούμε και όπως ε, γνωρίζετε έχουμε τρεις γνωμοδοτήσεις και τρει ε, εισηγητές. εξ αυτών βρίσκεται εδώ ο ίδιος αυτοπροσώπο, ο κ. Χριστιαν Έλερ, που είναι ο υπεύθυνο για το Horizon Ευρώπη. έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο, Επίτροπε. Νομίζω ότι και ο κόσμος και το Κοινοβούλιο ε, θεωρούν ότι είναι καινοτόμα αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι με τι πολιτικά μέσα θα πετύχουμε το στόχο μας. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε προς την σωστή κατεύθυνση και έτσι είναι το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να επιτύξετε φιλοδοξία. Έχουμε μελετήσει αυτά τα οποία έχετε δημοσιοποιήσει όσον αφορά τα του προπολογισμού και αυτά τα 160 εκατομμύρια τα οποία ε, επισημάνατε ως ε, πρικοδότηση που θα βοηθήσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο δεν θα θέλαμε να πάει χαμένο. Είναι σημαντικό επομένω. Για τον προϋπολογισμό τώρα, δύο ερωτήματα. Λόγω των ιστορικών διαπραγματεύσεων δίνεται η εντύπωση ότι έχουμε 10 δις που θα πάνε στην Γεωργία. Εντάξει, μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Αλλά είναι η γεωργία η προτεραιότητα όσον αφορά την έρευνα. Πάντως, θα έφερνε σε μηχανία πολλούς αυτό το μήνυμα. Επίσης, να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, το οποίο είναι σημαντικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και έχουμε άλλα 3,5 δις, τα οποία αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα. Και αυτό θα αποτελέσει πολιτικό πρόβλημα. Για τα άλλα ζητήματα τώρα, Και εμείς θέλουμε διεύρυνση στο Κοινοβούλιο και επίσης απλώς ουσίας να μάθουμε ακριβώς τι φιλοδοξίες έχετε, τι προοπτικές υπάρχουν. Τι είχε από το πρόγραμμα, τι προβλέπει ο προϋπολογισμός. Μήπως θα χρειαζόντουσαν περισσότερες αυξήσεις. Καλά έχουν γίνει κάποιες. Τώρα για το νέφος και τις πηγές open source, τις εφαρμογές open source στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε το fast track να, το, να επιμείνει περισσότερο και να είναι προσέγγιση από πάνω προς κάτω και όχι το αντίθετο. Επίσης, ε, μας είπατε για τις εταιρικές σχέσεις, για τις αποστολές, για το σχέδιο κειμένου που αναφέρεται στο στατικό προγραμματισμό που αφήνει να καταλάβουμε πώς θα έχει η διαδικασία και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί πάντως. Οπότε, το σημαντικό είναι να έχουμε εδώ πέρα ένα μείγμα συνέχειας και φιλοδοκίας και για τι εταιρικέ σχέσει να έχουμε κάποια παραδείγματα μίμηση, όπω το Clean το οποίο είναι παράδειγμα μίμηση για όλο τον κόσμο. Θα επανελευθεί αυτή η επιτυχία. Επίσης, μας μίλησατε για τις ε, συνέργειες. Αλλά τι θα γίνει με τα διορθωτικά ταμεία, θα υπάρξουν συνέργειες. Πού θα τις βρούμε. Τώρα τελευταίο που καίει το κοινοβούλιο είναι το θέμα της ισότητας των φύλων. Είμαστε οι 82 Δεύτερη. αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την κατάταξη. Αλλά ακόμα 60.000 μηχανικοί που ασχολούνται με την έρευνα φεύγουν από την Ευρώπη. Υπάρχει όμως και αυτό το, το, το, το ποιοτικό στοιχείο το ηθικό στοιχείο για την στρατηγική, για την ισότητα των φίλων. Οι γυναίκες μετά από μια πενταετία το εν τρίτον φεύγει. 300.000 ευρώ κοστίζει η εκπαίδευσή τους. Πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουν και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους. Μην έχουμε δημοκρατικό πρόβλημα. Έχουμε πολλά θέματα, ε, συγγνώμη που σας τα είπα βιαστικά, ακόμα διαβάζονται τα ζητήματα αυτά τα κείμενα του συναδέλφου, αλλά αν μπορείτε να σταθείτε για να μα τα φωτίσετε αυτά τα σημεία. Ευχαριστούμε, συναδέλφοι. Ο κύριος Ντανίκα έχει ασχοληθεί με το Horizon Europe, το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. Ο, κύριο κύριος Καμπεθόν Ρουίθ θα τον αντικαταστήσει και εκ μέρους του Ντάν θα μας πει δύο λόγια ως παρατηρήσεις του. Ευχαριστώ. Λέει κύριε Καπιθονορή. Ναι και με την ε, ευκαιρία να παρέμβω κι εγώ. Να μην ξενιτήσω το λόγο για να πω τα δικά μου. Τέλος, απ'λευράς του κυρίου Νίκα. Ζητεί να σας πω τα εξή. Τονίζεται τα εξή εταιρεία ότι χρειάζεται πιο φιλόδοξος προϋπολογισμός. Ξέρουμε ποια είναι τα ποσά προβλέπονται και το Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει την υπόθεση θέλει να αυξηθεί η για να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει. Επίσης, ζητεί να προωθήσουμε μία δίκαιη κατανομή σε όλες τις ομάδες της ερευνητικές στην Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα να είναι παραγωγικό, να είναι θετικό, να προσφέρει προστιθεμένη αξία. Και έτσι να ωφεληθεί η κοινωνία και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω. Χρειάζεται αύξηση του προϋπολογισμού, όπως τα έχει πει το Κοινοβούλιο στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Μας προβληματίζουν αυτά που λέει η Επιτροπή. Γιατί για δεύτερο και τρίτο πυλώνα οκ, αλλά στον πρώτο πυλώνα δεν βλέπουμε καμία αύξηση. Τι θα γίνει με την αριστεία. Πολύ σημαντικό να υπάρχει αναλογική αύξηση παντού. Παναλαμβάνω, προβληματίζομαι τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Θα πρέπει το πρόγραμμα να έχει πιο εγκάρσιο χαρακτήρα όσον αφορά το δεύτερο άξονα γιατί οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να επιστρατευτούν. Και να υπάρχει τέτοιο πνεύμα, τέτοια λογική που να μην υπερισχύει το ένα μέτωπο, ένα τομέα, ένα άξονα εναντί άλλου. Τελικά τι θα καθισχύσει το, η ποιότητα του κάθε προγράμματος ή άλλη μεταβλητή. Θα πρέπει πάντως να υπάρχει μια επιτροπή προγράμματος αν άξονα. Και όσον αφορά αυτού του είδους την μπλε αύξηση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τους άξονες στο μέλλον, ούτως ώστε να υπάρχει μια σύμπραξη τέτοια μπλε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. και μπορείς να έχουμε συνέργεια μέσω αυτή τη ιδιωτική χρηματοδότηση. Τώρα για την υγεία. Να καλύψουμε ένα εκατομμύριο Ιδιωμάτων. Και έτσι να φροντίσουμε να μην παραβλαβεί ο προϋπολογισμός να δούμε συγκεκριμένα τι θα γίνει με τις ε, αποστολές και όσον αφορά τις ΜΜΕ, το σχετικό εργαλείο είναι πάρα πολύ θετικό. Να δούμε τι θα γίνει στην τρίτη φάση, τι θα γίνει από την προβλεψιμότητα και την αξιοπιστία, σημαντικά. Όπως είπατε πρόεδρε, πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τη χρηματοδότηση. Οι ΜΜΕ εξαρτώνται κατά πολύ από τις ενισχύσεις, περισσότερο από ό,τι από τη δανειοδότηση. Να φροντίσουμε να συμμετάσχουν οι ΜΜΕ. Οπότε ανησυχώ γιατί θα πρέπει να διατηρηθούν οι προβλέψεις για τις ιδιορυθμίες του προγράμματος. Δεν έχω καμία αντίρρηση για κάποιες χώρες που έχουν πρόβλημα να ληφθεί αυτό υπόψη αλλά για την αναθεώρηση του προγράμματος επίσης να υπόψη κάποιες χώρες που δεν το χρειάζονται το πρόγραμμα όπως το Λουξεμβούργο και το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 προβλέπει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάποιες συγκεκριμένες χώρες ή περιφέρειες. Άρα, να δούμε και σε αυτή την περίπτωση ποιες περιφέρειες έχουν πρόβλημα συμμετοχής. Πολύ ενδιαφέροντας που μας είπατε για την συνέργεια. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αξιοποιήσουν περισσότερο τους πόρους. Να μην επισέλθουμε τώρα στις λεπτομέρειες, αλλά έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα υποβάλω τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, κλείνω, κλείνω, Πρόεδρε περισσότερο φιλόδοξη για την ισότητα ανδρών και γυναικών και επίσης για στην, να ε, έχουμε αυτού του είδους την αποσύνδεση όπως προβλέπει η ενδιάμεση αξιολογησία, και στην ε, έρευνα να έχουμε ισότητα στην ε, συμμετοχή και θετικά τόσο πολύ για τις εταιρικές σχέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής τώρα. για το ECR, του Σενόφσκι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τον Επίτροπο Μέδες ε, που έρχεται για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή, ΤΡΕ, για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι η χρηματοδότηση της επιστήμης, ε, της καινοτομίας και της έρευνας στο μέλλον. Συμφωνώ ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη, την ατμομηχανή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και εγώ και ως μέλος ε, της Επιτροπής ΤΟΑ ήμουν ανέκαθεν ε, θερμός υπέρμαχος της έρευνας και της καινοτομίας και χαίρομαι για την αύξηση των κονδυλίων. Γιατί η έρευνα και η καινοτομία θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Κάτι που θα επηρεάσει και το μέλλον μας στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες, Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να μιμούμαστε τυφλά ή να αντιγράφουμε το αμερικανικό σύστημα. Γιατί το αμερικανικό σύστημα δημιουργήθηκε υπό άλλους όρους και συνθήκες και ακολούθησε και διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Πάντως θα πρέπει να στηρίξουμε τις δικές μας νεοφυείς επιχειρήσεις πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο. Τι είδου κεφάλαια κινδύνου θα στηρίξετε για τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί τέτοια venture capital θα πρέπει να έχουν πιο κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε διαφορετικά τους κινδύνους και διαφορετικά τους αξιολογούμε. και μερικές φορές δεν είμαστε τόσο ε, ενθουσιώδης υπέρμαχοι του επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου κινδύνου, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τέτοιο κεφάλαιο χρειάζεται για να στηρίξει την έρευνα και την ε, καινοτομία στην Ευρώπη, venture capital. Δεν κατάλαβα πώς ε, από το έγγραφό σας θα αντισταθμίσουμε τους κινδύνους του επιχειρηματικού κεφαλαίου, του επισφαλούς κεφαλαίου, ώστε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα την έρευνα και την καινοτομία. Μας ε, υποσχεθήκατε αύξηση αρκετών προγραμμάτων, κάτι που θα είναι δύσκολο στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Πάντως η, και η δική μου πολιτική ομάδα είναι υπέρ της αύξησης των σχετικών κονδύλιων, παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις που έχουμε για άλλα προγράμματα. Κύριε Βιέριν από την Άλντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω που προσήλθατε για να φωτίσετε τις ερωτήσεις που έχουμε για τον ορίζοντα Ευρώπη. Όπως και οι συνάδελφοί μου, έχω πολλές ερωτήσεις. Για την ώρα, ωστόσο, θέλω να τονίσω ιδιαίτερος μία. Θα ήθελα, δηλαδή, να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ποια θα είναι η ισορροπία μεταξύ των πρωτοπόρων προγραμμάτων και των επιταχυντών. Ε, αναφέρομαι στην κατανομή κονδυλίων, αλλά και στην στόχευση και των δύο αυτών ε, project. Και θέλω να μιλήσουμε ακόμα και για τις ε, κοινοπραξίες. Υπάρχει ακόμα μεγάλη βεβαιότητα σχετικά, αλλά είμαι βεβαίο ότι μπορείτε να εξηγήσετε πότε θα πρέπει, πότε θα έχουμε ένα ξεκάθαρο σήμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον των κοινοπραξιών. Και τέλος, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης ε, Ευρω... Ε, Horizon Ευρώπη και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαι βεβαίω ότι θα ξαναειδωθούμε για να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά περισσότερο. Πρώτος σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. για τον ε, συνοπτικό τρόπο με τον οποίο θέσατε ξεκάθαρα τα θέματα σας. Ο κύριος Νταλούντερ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την ε, καλή πρόταση και βέβαια υπό τις δυσχερείς ε, περιστάσεις μπορούμε να είμαστε περήφανοι για πολλά τμήματα της προτάσεως. Χαίρομαι που βάζουν την, ε, την αριστεία στην, στο προσκήνιο. Έχω τώρα τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, δράση υπέρ του κλίματος. Έχοντας υπόψη τον έλεγχο που έγινε για τον ορίζοντα 2020, είδαμε ότι δεν εκπλήρωσε τους στόχους του, που ήταν 35% και θα καταλήξουμε μονάχα στο 30%. Και ο έλεγχος επίσης αμφισβητεί εάν τα 37% είναι επαρκή σε ό,τι αφορά ένα project το οποίο ε, έφερε το τίτλο Climate Action, τελικώς δεν ήταν. Τώρα, ρωτώ, ποια έχει έγκυα... Ε, δίνεται για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθεί το 35% στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Δεύτερο, με αυτό το ρυθμό over subscription που βλέπουμε, τι κάνει εκ παραλίλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι θα συμβάλλουν με το 3% οι χώρες μέλη που είναι ο στόχος σύμφωνα με τη διακήρυξη της Βαρκελόνης. Τρίτο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούν να επιταχύνουν. Το Συμβούλιο όμως φαίνεται να κολλησιεργεί. Ερώτηση. Τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία ώστε να δούμε να αποδίδουν οι προτάσεις ίδια το 2021. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης της Ενωτικής Αριστεράς. Πρόεδρε, ε, θα, ήθελα και εγώ εκ μέρους της Γκουέτζιερ να καλωσορίσω τον Επίτροπο έδα, εδώ και για την παρουσία που έχει κάνει. Θέλω να πω, κύριε Επίτροπε, ότι μιλήσατε στην αρχή για επανάληψη. Βεβαίω, μοιραία και εμεί επαναλαμβανόμαστε στην κριτική που ασκούμε σε σχέση με τα προγράμματα και το τι εφαρμόζεται. Να πω ότι το νέο πρόγραμμα Ορίζοντα έχει θετικά στοιχεία, αλλά κατά την άποψή μα έχει και πολλέ αδυναμίε που πρέπει να διορθωθούν. Αρχικά, εμεί εκτιμούμε ότι οι συνέργειε μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιωτικού τομέα ε, που ευνοούνται από το πρόγραμμα μετατρέπουν πολλές φορές την έρευνα σε εργαλείο των μεγάλων εταιριών σε βάρος της κοινωνίας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το σημειώσουμε. Ε, το οποίο γιατί οι πολυεθνικές εταιρείε πάντοτε βλέπουν τα πάντα στη βάση των δικών του στενών ιδιαίτερων συμφερόντων. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι να δοθεί έμφαση για να συνέρευνα για την εξυπηρέτηση των αγκών της κοινωνίας. Βεβαίω, αναμένουμε ότι μέσα από τη συζήτηση και τη δική μας πίεση στο Ευρωκοινοβούλιο θα αυξηθεί το διαθέσιμο κονδύλι ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα και νομίζω ότι είναι ένα σημείο εδώ που συμφωνούμε ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Επίση, ε, ω ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, έχουμε ξεκάθαρη θέση ενάντια στην πρόταση για χρηματοδότηση τη έρευνα στο στρατιωτικό τομέα Κατά την άποψή μα αυτό οδηγεί στην περαιτέρω στατικοποίηση τη Ένωση με καταστροφικά αποτελέσματα για του λαού, το είπαμε πολλέ φορέ. Επίση, θέλω να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματο Ορίζοντα 2020, δυστυχώ χρηματοδοτούνται φορεί που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο μερικέ φορέ. Αναφέρομαι σε φορεί του Ισραήλ, οι οποίοι ε, δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το εξετάσετε με πολύ σοβαρότητα. Χρειάζεται επίσης να προωθήσουμε ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις, ώστε το πρόγραμμα να προωθεί την έρευνα για στήριξη πρώτη στάδης πραγματική οικονομία για κοινωνική ανάπτυξη και ε, δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία. Τέλο, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν ισότιμη πρόσβαση. Γιατί δηλαδή, είναι αλήθεια σήμερα δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη ισότιμη πρόσβαση στα προγράμματα. Και πώ θα στηριχτούν ιδιαίτερα οι πολύ μικρέ και μικρόμεσε επιχειρήσει, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα ε, να αξιοποιήσουν ακριβώ τα προγράμματα, να έχουν πρόσβαση, για να μπορέσουν να συμμετέχουν ισότιμα και να αξιοποιήσουν όλε τι δυνατότητε που δίνουν τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ κυρία Κάπελ από το ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς και Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για την καλή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας θεωρώ υπόδειγμα ε, συνεργασίας με τους Ευρωβουλευτές και πάντοτε είστε διαθέσιμος για ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τη σημερινή συζήτηση μου φαίνονται τρία πράγματα, ιδίω από τη σκοπιά των επιχειρήσεων, ότι έχουν μεγάλη σημασία. Πρώτον, ότι για την καινοτομία και έρευνα αυξάνονται τα κονδύλια σε, στα 100 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση, εξακολουθούν είναι λίγα, αλλά έχει συμβολική αξία το γεγονός ότι ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας λαμβάνουν μεγαλύτερη αξία, διότι είναι βέβαια και σημαντικός μοχλός για την απασχόληση στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, βρίσκω θετικό αυτό που είπατε σήμερα, ότι για να συμμετέχουν στο ε, Horizon Europe μπορεί να υπάρξει συγχρηματοδότηση και από τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό το ζητούμε από καιρό και είναι σημαντικό για να χρησιμοποιηθούν και τα κονδύλια των διαθετικών ταμείων συγχωρισμένοι. Επίσης, πολλά χρόνια συζητείται κάτι, ανεπιτυχώς όμως, περισσότερα κονδύλια να επενδυθούν για την διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων και όχι μόνο για την έρευνα βάση. Τώρα έχω δύο σύντομες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσει. Το ένα για το Horizon Europe που είναι σημαντική, είναι μεγάλη σημασία του προγράμματος και στη χώρα μου την Αυστρία 460 επιχειρήσεις έλαβαν χρήματα από το Horizon Europe με συνολικό ποσό 23 εκατομμύρια και βρίσκω πολύ σημαντικό να παραμείνετε στους τρεις πυλώνες και έβεβαιος ε, αύξηση των κονδυλίων αλλά στο Horizon Europe θα περιλάβετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δέσμευση κονδυλίων της τάξη του 20%. Θα το ξαναδούμε δηλαδή στο νέο ΠΔΠ. Και όπως ήταν έω τώρα θα συνεχίσει το πρόγραμμα να αξιολογείται διαρκώ και να προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών. Και τέλος το market program. Και εδώ είναι θετικέ οι εμπειρίες από τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Και ρωτώ ποιο θα είναι εδώ ο προσανατολισμό. Εάν δηλαδή θα ενισχύσετε το Enterprise Europe Networking ή θα κινηθείτε προς την κατεύθυνση περισσότερη προστασία των καταναλωτών ή και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις σας. Αυτοί ήταν οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων και οι εισηγητές βέβαια. Τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, ο κύριος Μαρτέλ, Μαρτέν, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Τα είπαν κάπως γενικότερα. Οι συνάδελφοί μου, εγώ έχω κάτι πιο στοχευμένο, έστω και αν δεν είναι απολύτω θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά περισσότερο κύριο Σεύκοβιτς, αλλά και εσείς είστε αφεντικό εκεί στην έρευνα, δηλαδή για την Airbus. Airbus. για την συνεργασία στην έρευνα που είναι απολύτως απαραίτητη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι Κινέζοι προχωρούν σε μαζικές επενδύσεις, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν τι είδους κονδύλια μπορούν να ενισχύσουν την έρευνα, την καινοτομία κλπ. Θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να υπάρχει δηλαδή ένα ιδιαίτερο προπολογισμό εν ώψη και των προσανατολισμών που θέτουμε, δηλαδή να περάσει η αυτοκίνηση σε ηλεκτροκίνηση και να τηρηθούν ποια είναι τα σφάλματα του παρελθόντος, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά τόξα. Μπορείτε να δώσετε λοιπόν τα σχετικά κίνητρα που είναι αναγκαία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να καλωσορίσω και εγώ τον Επίτροπο, τον κύριο Μοέντα, στην Επιτροπή μας και ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας ότι προφανώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομία είναι κάτι πολύ σημαντικό και θεωρώ σημαντική την πρωτοβουλία σας, όπως επίσης το ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα παραδείγματα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980 με την Bay Doll Act υπάρχει αυτό που λέγεται προτίμηση για τη βιομηχανία των ΗΠΑ, δηλαδή Preference for United States Industry. Και επομένως οι ευρυσιτεχνίες και οι πατέντες, οι οποίες διαμορφώνονται με δημόσια κονδύλια των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει δέσμευση από τις επιχειρήσεις να αξιοποιούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνο κατ' εξαίρεση να μπορούν να αξιοποιούνται από επιχειρήσεις εκτός ΗΠΑ. Επειδή και η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι πλέον αφελής, αλλά τα κονδύλια τα οποία επενδύουμε τα δημόσια κονδύλια για τη δημιουργία τεχνίας και πατέντας πρέπει να διασφαλίσουμε να αξιοποιούνται από τις ευρωπαϊκές επιχείρησεις εντός της Ευρώπης και μόνο κατ' εξαίρεση να μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης. Μήπως ήρθε η ώρα αυτό το καλό παράδειγμα των ΗΠΑ που προστατεύουν τα δικά τους χρήματα, τις δικές τους επενδύσεις, τη δικιά τους προστιθέμενη αξία να την αξιοποιήσουμε και στην Ευρώπη. Να μην πληρώνουμε δηλαδή κεφάλαια για να έχουμε έρευνα, να έχουμε καινοτομία, να έχουμε βρυσιτεχνίες και στο τέλος αυτές να αξιοποιούνται τσάμπα θα έλεγα από επιχειρήσεις κινέζικες ή αμερικανικές να αξιοποιούνται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και θα ήθελα αυτό να το δείτε γιατί η εμπειρία σας είναι γνωστή. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που δίνουν εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες ως παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, colleague. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόχλιτσεκ, ο αντιπρόεδρός μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα και εγώ να κάνω λίγα σχόλια. Με βλέπετε. Ε, λίγα σχόλια. Αν σας δημιουργεί πρόβλημα το ότι μιλάω τσεχικά, μπορώ να μιλήσω και άλλη γλώσσα, με αποτιμάτε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό του προϋπολογισμού ε, του ΑΕΠ που αφιερώνεται στην έρευνα. Γιατί έχουμε θέσει στόχο 3%. Αλλά δεν το καταφέρνουμε σε όλες τις χώρες, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αναφερθήκατε σε κλάστερ. Αυτά τα κλάστερ θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλους, όχι μόνο στις ε, πιο ισχυρές χώρες, ή πιο εύπορες. Θα πρέπει και οι μικρομεσαίες χώρες να μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοια κλάστερς. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις μικρομεσαίες χώρες. Τώρα, για τη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα καταλήγει σε λίγα διπλώματα ευρυστεχνίας. Σημαντικά όμως είναι έστω και αυτά τα λίγα διπλώματα ευρυστεχνίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα clusters. Ίσως είμαστε επικεντρωμένοι στην εφαρμογή, αγνοώντας κάπως ή αδιαφορώντας κάπως για τη βασική έρευνα. Τρίτο σχόλιο. Τεχνικά επαγγέλματα και πόσο ελκυστικά είναι. Η Ευρώπη τον προηγούμενο αιώνα ήταν γνωστή για την παραγωγή έγκριτων εμπειρογνωμόνων και ειδικών. Σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι η μηχανική και άλλα τεχνικά επαγγέλματα λείπουν από την Ευρώπη. Υπάρχει ένα έλλειμμα τέτοιων τεχνικών επαγγελμάτων. Εκεί που παλιά είχαμε 100 αποφύτου τεχνικών ε, πανεπιστήμιων και σχολών, τώρα έχουμε 20-30. Και τέλος, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απαλλάξουμε την οικονομία μας από τον άνθρακα. Αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε υπερβολικά άλματα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο υδρογόνο. Να ξεκινήσουμε με την ηλεκτρόλυση, με την αποθήκευση και με κάποιες ενδιάμεσες φάσεις μέχρι να βελτιώσουμε τεχνικά τις κυψέλες υδρογόνου. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες έρευνες εκεί, αλλά όχι αρκετές. Και έχουμε συμφωνήσει ότι 1% της ενέργειας μας θα πρέπει να προέρχεται από το υδρογόνο μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Τελευταία μιλήτρια στο κατάλογο είναι η κυρία Γκρίχερ. Τελευταία, αλλά όχι και λιγότερο σημαντική. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Κάρλος Μοέντας που ξαναήρθε στην Ήτρε, γιατί έχουμε πολύ επικοδομητικό διάλογο και με σας και με το επιτελείο σας από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Και θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με τον φίλο από τους Πράσινους και να στενιστώ τα σχόλια που ακούσαμε για την ηλεκτροκίνηση. Όπως είπαμε και στην τελευταία μας συνεδρίαση, το Brexit ε, θα είναι αμοιβαίως αρνητικό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στην καινοτομία και την έρευνα. Θέλουμε να πρωτοστατούμε στην Ευρώπη, στην ενέργεια, στην ψηφιακή οικονομία, στις ενέργειες και στις θέσεις απασχόλησης και την ε, οικονομική ανάπτυξη και χαίρομαι που ήταν θετικό το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου της περασμένης εβδομάδας. Θα πρέπει όμως να επενδύουμε σε όλες τις αλυσίδε της παραγωγής και στη διάδοση και την αξιολόγηση. Γιατί κατά παράδοση επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην παραγωγή και όχι αρκετά, κατά τη γνώμη μου, στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και μετά στη διάδοση της γνώσης και στην αξιολόγηση. Κάποιοι μίλησαν για την ισότητα και την των φύλων. Όντω, εκεί έχουμε κάποιες, θα πρέπει να κάνουμε κάποιε βελτιώσει. Και ίσω ε, εσύ καλώ θα μπορούσε να δώσει την απάντηση που δεν μπορεί να δώσει η Βρετανική κυβέρνηση μέχρι στιγμή. Ποιο θα είναι ο ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλα αυτά τα πανέμορφα πράγματα και τι προτάσει σα. Ευχαριστώ. Ελπίζω να λάβετε μια ξεκάθαρη απάντηση και εσεί από τον Επίτροπο αργότερα και ευχαριστώ θερμά του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στη συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν μα έχει μείνει και πολλής χρόνος, γι' αυτό και θα πρέπει να οργανωθούμε άρτια για να μπορέσουμε να τα διεκπαιρεώσουμε όλα μέσα σε ένα οκτάμινο. Κάτι που δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αλλά θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να ετοιμαστούμε για αυτό. Πολύ σημαντικός και ο διαρθρωμένος διάλογος, γιατί χάρη σε αυτόν θα μπορέσουμε να διεκπεράσουμε αυτά τα θέματα το επόμενο οχτάμινο και με την επόμενη Προεδρία, τη Ρουμανική. Καλώς έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά το, τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για τις ερωτήσεις τους, για τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ και για όλες τις επαφές που είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και τις συζητήσεις. Θα ξεκινήσω με τα σχόλια του Κρίστιαν Έλλερ. Και την πρώτη ερώτηση που αφορούσε το δημοσιονομικό, τον προπολογισμό. Με ρώτησε αν είμαι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα. Είπα ναι. Αν αρκεί, θα έλεγα όχι. Αλλά αυτό έχουμε. Με αυτό θα πορευτούμε. Και χαίρομαι πάντως που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη μάχη του. Και ξέρετε σε ποιο, σε ποιο το πλευρό είμαι σε αυτή τη συζήτηση. Πάντως το επίτευγμα μέχρι στιγμής είναι σημαντικό. Με ρωτήσατε και για το θέμα τρόφιμα και φυσική πόρη. Είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση του σημείου αυτού του προϋπολογισμού, του τομέα αυτού του προϋπολογισμού, γιατί προηγουμένως ήταν πολύ πενιχρό το σχετικό κονδύλιο. Και αν δούμε άλλα κλάστερ, όπως το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα, εκεί βάλαμε 15 δισεκατομμύρια. Η ψηφιακή, ψηφιακός κλάδος 15 δισεκατομμύρια. Είπαμε όμως, αν το μέλλον ανήκει στην ε, ψηφιακή βιομηχανία και βάζουμε εκεί 15 δισεκατομμύρια ή για, το, για την ενέργεια, το κλίμα και την κινητικότητα και βάζουμε και εκεί 15 δισεκατομμύρια και αν μιλούμε για τους φυσικούς πόρους, την κυκλική οικονομία, για το τι θα φάμε, πώς θα τραφούμε στο μέλλον. Αυτό είναι το παν. Οπότε ακόμη και αν ε, το θεωρείται μεγάλη αύξηση, νομίζω ότι ήταν απολύτω απαραίτητη αυτή η αύξηση σε αυτό το κλάστερ των τροφίμων και των φυσικών πόρων. Γιατί στο παρελθόν υστερούσε. Και είμαι υπερήφανο για την ε, δραστική αυτή αύξηση, γιατί πραγματικά δείχνει τι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τομέα αυτό. Και γι' αυτό σας ε, έδωσα και τις σχετικές εξηγήσεις για τα προτινόμενα από ποσά. Επίσης, μιλήσατε για την διεύρυνση, το widening, τη διεύρυνση και την ε, κοινή ε, αξιοποίηση της αριστείας. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε τώρα, το widening, της διεύρυνσης. Ήταν θέμα αρχής να διπλασιάσουμε αυτό το σκέλος του προγράμματος, κάτι που είναι απαραίτητο για πάρα πολλές χώρες και γι' αυτό θα σταθούμε σε αυτό αυτή τη θέση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από εκείνο το πεδίο εφαρμογή. Επίση, μιλήσατε για το νέφο, την εφολυπολογιστική και το νέφο τη ανοιχτή επιστήμη. περνάμε πια από τα λόγια στα έργα. Και αυτό το νέφος της επιστήμης, το Science Cloud, θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα, να περάσουμε στον οδικό χάρτη, να ξέρουμε τι θέλουμε και σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Και υποβάλλατε και ένα πιο τεχνικό ερώτημα για την ιδέα του στρατηγικού προγραμματισμού ή του στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Θα ήθελα να είμαι σαφές ότι αυτή η ιδέα του στρατηγικού προγραμματισμού προϋπήρχε και είναι πολύ σημαντικό ε, περνά, περνώντας από τα νομικά έγγραφα στο πρόγραμμα εργασιών και προς το στρατηγικό σχεδιασμό. Και ίσως αυτή τη φορά σταθήκαμε πιο εκτενώς αυτό λόγω των αποστολών και της σημασίας των αποστολών. Γιατί θα χρειαστεί να προσδιορίσουμε τις αποστολές βάσει κριτηρίων που θα πρέπει να προσυμφωνηθούν. Πάντως, σημειώνω την παρατήρησή σας για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ίσως εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο σαφείς και θα το κάνουμε στο μέλλον για να δούμε ποια, τι μορφή θα έχει ο στρατηγικός σχεδιασμός, τι θα είναι και τι δεν θα είναι, αυτή τη φορά μιλήσαμε λίγο πιο ε, διεξοδικά για τον στρατηγικό σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά τις συνέργειες, ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Νομίζω ότι η διατύπωση θα περιληφθεί στο πρόγραμμα για τα διαρθρωτικά ταμεία. Στην πρότασή μας δεν είχε τόσες λεπτομέρειες. Το πρόγραμμα για τα διαρθρωτικά ταμεία περιείχε τις λεπτομέρειες της πρότασης. Εκεί θα περιληφθεί γιατί ίσως δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα όπως το επισήμανε πολύ εύστοχο ο κύριος Έλλερ. Δηλαδή, περιέγραψα κάτι που δεν ε, αναφέρεται σχολαστικά στην πρόταση. Υπάρχει όμως, υπάρχει στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά στα διαρθρωτικά ταμεία. Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, το επισήμαναν η Σολεδάδη, η Τερέζα και άλλα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Σε ό,τι αφορά το φύλλο, την ισότητα των φύλων, η σημαντική συζήτηση που θα συνεχιστεί και στο μέλλον είναι ότι γνωρίζουμε ε, πώς έχουν λειτουργήσει οι πολιτικές ισότητα των φύλων στις, στις σκανδιναβικές χώρες. Και ξέρουμε ότι οι πολιτικές αυτές λειτουργούν όταν τις προωθούμε, όταν τις, τις εμπλουτίζουμε με στόχους, όταν τις προωθούμε. Νομίζω ότι έχει γίνει σημαντικό έργο μέχρι στιγμής, έχει σημειωθεί πρόοδος και πολλές γυναίκες επιστήμονες έρχονται στα σεμινάρια μας και στα πάνελ μας και μου λένε ότι νιώθουν πολύ οικία γιατί έχουμε ποσοστό γυναικών 30 με 40% στα πάνελ μας. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε δεν θα πρέπει να μαστιγωνόμαστε συνέχεια και να είμαστε τόσο επικριτική, γιατί πραγματικά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο θέμα τη ισότητα των φύλων. Φυσικά, εξακολουθούμε να είμαστε φιλόδοξοι και σα διαβεβαιώ ότι εστερνίζομαι αυτή την ανάγκη και τη φιλοδοξία. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια τη Σολεντάτ και του Νταν Νίκα. Θα σας μιλήσω ισπανοπορτογαλικά, Σολεδάδ. Καταρχήν, για τον προϋπολογισμό. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αν και θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο φιλόδοξοι. Αλλά ελπίζω να βρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμάχους για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να αντιληφθούν οι χώρες την ανάγκη αυτού του προπολογισμού. Και θεωρώ ότι το 100 είναι πολύ συμβολικό νούμερο. Και ακριβώ επειδή είναι συμβολικό ο αριθμό το 100, ελπίζω να αντιληφθούν και οι χώρε το συμβολισμό που έχει αυτό το νούμερο το 100. Όταν η μίλησε για την ηθαγένεια. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γι' αυτό και οι αποστολές είναι πολύ σημαντικές, γιατί οι αποστολές επιστήμης ακριβώς ε, θέλουν να εμπλέξουν και τους πολίτες. Και επίσης, ε, για να συμμετέχουν οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν ότι το ζήτημα τους μιλάει, το τομέα τους μιλάει και αυτό θα πρέπει ε, να κάνουμε στο μέλλον, να εξηγήσουμε καλύτερα τις δράσεις μας. Και αυτό θα το κάνουμε μέσω των αποστολών. Επίσης, με ρωτήσατε για τον πρώτο πυλώνα και τις αυξήσεις. Αν ε, εξετάσετε όλες τις δημοσιονομικές γραμμές του προϋπολογισμού και δείτε ποιο είναι το πιο σημαντικό κονδύλιο. Το πιο σημαντικό κονδύλιο είναι αυτό που αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία. Ε, έρευνα, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Φροντίσαμε ε, το πιο μεγάλο ποσό που έχουμε από όλο το πρόγραμμα να είναι από τον πρώτο πυλώνα. Και φυσικά είναι δύσκολο να κάνουμε επιλογές, αλλά επιλέξαμε να δώσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό το το μεγαλύτερο ποσό στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Αυτό για μας ήταν θεμελιώδες. Επίσης, ε, μας μιλήσατε για την κοινωνική πρόκληση. Το, η κοινωνική πρόκληση και η πρόκληση των κοινωνικών επιστημών είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Και αν ρίξετε μια ματιά στην πρότασή μας, και την εξετάσετε πιο προσεκτικά θα διαπιστώσετε ότι ακριβώς έχουμε κάποιους τομείς παρέμβασης γιατί λέμε ότι είναι σημαντικό να συμβάλλουν οι κοινωνικές επιστήμες για να προσπίσουμε τη δημοκρατία. Και θέλουμε περισσότερα σχετικά προγράμματα. Επίσης, πολιτιστική κληρονομιά, ε, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ε, κοινωνική ανθεκτικότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να ε, προσδιοριστούν με σαφήνεια και να βρίσκονται σε όλο το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα. Και αυτό το τμήμα των κοινωνικών προκλήσεων... Α, ήδη έχει έρθει η Επίτροπος και περιμένει. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία αφορά ακριβώ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και θα συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία ω επιταχυντή για το μηχανισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα βελτιωθεί. Και το fast track για την καινοτομία επίση θα βελτιωθεί. Δεν θα διαγραφεί. Με πιέζει αρκετά ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να απαντήσω σε όλους και θέλετε στη συνέχεια και διμερώς να συζητήσουμε. Ο κύριος Στοσενόφσκι με ρώτησε για το κεφάλαιο κινδύνου, το venture capital. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εγώ είμαι θερμός υπέρμαχος της αύξησης του κεφαλαίου κινδύνου και έχουμε πια το Ταμείο των Ταμείων, Fund on Funds. Ένα ευρώ από δημόσια κονδύλια να λαμβάνουμε τρία ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα. Και τώρα έχουμε μια επιλογή των υπευθύνων. Ήδη έχουμε υπογράψει το πρώτο συμβόλαιο με τον πρώτο υπεύθυνο. Θα πρέπει τώρα να βρούμε ιδιωτικά κεφάλαια. Και πριν από λίγες μέρες ήμουνα στην Πράγα και πραγματικά συναρπάστηκα από την έντονη επιχειρηματικότητα και ευρηματικότητα που βρήκα εκεί. Ε, κυρία Τελίντε, με ρώτησε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το πρωτοπόρα προγράμματα και τους επιταχυντές. Στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβουλίο δεν θα προσδιορίσουμε αμέσως τα ποσά. Θα γίνει με προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Πάντως, οι μικρομεσαίες επιχείρησεις που θα είναι στο Fast Track θα μπουν στον επιταχυντή βλέπετε έτσι την κατανομή μεταξύ των διαφόρων σταδίων από το Pathfinder μέχρι τον επιταχυντή. Ο κύριος Λαλούντε ε, ρώτησε σημαντικά θέματα για την κλιματική δράση. Ο στόχος δεν ε, έχει εξαλειφθεί, διατηρείται. Η ερώτησή σας όμως ήταν πιο δύσκολη. Με ρωτήσατε τι συνέβη, γιατί δεν έχουμε υλοποιήσει το στόχο. Νομίζω ότι αυτό έγινε για διάφορου λόγου. Σω ένα ήταν ότι πολλοί από την έρευνά μα που γίνεται από την, κορυφή προ τη βάση, δεν, ε, από την βάση προς την κορυφή δεν ελήφθη υπόψη. Έχουμε σχέδια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου που ε, συνέβαλαν στην κλιματική δράση, αλλά επειδή ήταν bottom-up δεν συμπεριλήθηκαν. Οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και θα πρέπει σίγουρα να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας και να έχουμε και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες όπως είπατε, γιατί το πιστεύουμε πραγματικά. Δεν θέλουμε απλώς να γίνουμε αρεστοί. Θέλουμε να υλοποιήσουμε το στόχο. Και για τις αποστολές σίγουρα θα έχουμε αποστολή και για το κλίμα. Επίσης μας μιλήσετε για το Συμβούλιο, μακάρι να έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προωθήσουμε τις θέσεις μας στο Συμβούλιο. Ο κύριος Ηλικιώτης με ρώτησε για τη μεταφορά μεταξύ ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών κύκλων. Είναι σημαντικό γι' αυτό ε, η ανοιχτή επιστήμη, τα ανοιχτά δεδομένα, η ανοιχτή πρόσβαση για όλα όσα είναι δημόσια. Γιατί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά. Να μην είναι ένα κλειστό κύκλωμα για τον ιδιωτικό τομέα. Να είναι ανοιχτά σε όλους, για κάθε ερευνητή, όπου και αν βρίσκεται στην Ευρώπη. Επίσης είπατε είστε κατά του στρατιωτικού σκέλους, αυτό όμω είναι εκτό συζήτηση, γιατί το ορίζον Ευρώπη αφορά το μη στρατιωτικό τομέα, το πολιτικό τομέα. Δεν έχει καμία σχέση με το στρατιωτικό τομέα. Οπότε εμεί αυτό το, το χαρακτηρισμό θα τον χαρακτηρίσουμε. Δεν ασχολούμαστε με στρατιωτική έρευνα στον ορίζοντα Ευρώπη. Σα διαβεβαιώ, μπορείτε να είστε ήσυχο γι' αυτό. Επίση, μιλήσατε για τι διαφορετικέ χώρε. Η επιστήμη είναι γέφυρα στι συγκρούσει. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλες τις χώρες, ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς που έχουμε, οι γέφυρες που μπορούμε να έχουμε με μια χώρα, με όποια χώρα και αν μιλάμε, και αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένα, όποια γέφυρα και αν έχουμε είναι σημαντική. Κυρία Κάπελ, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Και για τα καλά σας λόγια. Και νομίζω ότι οι συνεργασίες ε, στις οποίες αναφερθήκατε είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον διότι εν τέλει και τα διαρθρωτικά ταμεία και το Horizon Europe θα συνεργάζονται. Και όχι μόνο για τη βασική έρευνα, όπως είπατε. Μου μιλήσατε για το 20%, για το στόχο των 20%. Δεν υπάρχει στην πρόταση αυτή, αλλά εάν εξετάσετε το ιστορικό μας, θα δείτε ότι είχαμε υπερβεί το 20% υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαι βέβαιος ότι θα το διατηρήσουμε. Δεν έχουμε βάλει ωστόσο ρητά στόχο. Πολύ σωστά το παρατηρήσατε δεν περιλαμβάνεται διότι κατά τη γνώμη μου δεν μας χρειάζεται. Για τον κύριο Μαρτά με ρωτήσατε κύριε για κάτι που είναι σημαντικό. Η ιδέα, πώς να το πω τώρα στα γαλλικά, η ιδέα είναι για, για τους συσσωρευτές είναι ακριβώς αυτή. Αν έχει δηλαδή μια αποστολή η Ευρώπη που να λέει ότι οι Ευρωπαίοι φτιάξαμε ας πούμε ένα συσσωρευτή που θα επιτρέπει στα αεροσκάφη να πετούν ή ε, αυτοκίνητα ή ε, κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να το αντιληφθούν οι άνθρωποι αυτό. Εάν τώρα πείτε ότι ε, θέλουμε να φτιάξουμε τον καλύτερο συσσωρευτή, δεν ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, τι νοσπρόκειται. πρόκειται. Δηλαδή, για ποιο λόγο είπατε για τα 10 εκατομμύρια. Εγώ βλέπω, θα δούμε και στη συζήτηση μας μετά, ότι στη συζήτηση αυτή χρειάζονται, ε, χρειάζεται ένα είδος αποστολής. Για τον κύριο Μαριά, Νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην αμοιβαιότητα. Αντί να πούμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα πάντα, βεβαίω θέλουμε να προστατεύσουμε του πολίτε μα. Ο καλύτερο τρόπο για να προστατεύσουμε του πολίτε μα είναι να ζητήσουμε ε, να ε, λειτουργεί η αμοιβαιότητα. Αν λοιπόν το κάνω αυτό, εάν κάνω κάτι σε, για κάποιον και αυτό δεν το ανταποδώσει, τότε και εγώ δεν κάνω πιο δουλειέ με αυτόν. Ε, αμοιβαιότητα λοιπόν. Για τον κύριο Κόχλιτσεκ, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, πέρασα πρόσφατα από την Πράγα, μιλήσατε για διάφορα πράγματα, όπως τα τεχνικά επαγγέλματα. Παίρνω ένα που είναι σημαντικό, διότι δεν προλαβαίνω να σχολιάσω όλες αυτές τις παρατηρήσεις, τις οποίες δέχομαι βεβαίως, αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ελκυστικά τα τεχνικά επαγγέλματα. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντικά για τους νέους. Σημαντικά και ουσιώδη για τη ζωή τους. Εν πάντα στον ψηφιακό κόσμο θα πρέπει να εργαστεί κανείς στα επαγγέλματα αυτά. Και πρέπει να διασυνδεθούν οι διάφοροι κλάδοι, οι τέχνες με τα τεχνικά επαγγέλματα για να έχουν και πλάκα τα τεχνικά επαγγέλματα για να είναι τελικώ ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τα νέα παιδιά. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα προγράμματά μα λοιπόν για να γίνουν τα επαγγέλματα αυτά πολύ πιο ελκυστικά. Άκουσα δηλαδή το μήνυμά σα, έλαβα το μήνυμά σα τέλο για την Τερέζα, δεν μπορώ να απαντήσω για την Βρετανική κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές στην πρότασή μας ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και είναι τόσο ξεκάθαρο στην πρόταση που τώρα αναμένω την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι θεωρώ ότι αυτά που βλέπουμε με τις συνδέσεις με τις τρίτες χώρες όπως ζήτησε το Συμβουλίο είναι κάτι ξεκάθαρο και κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον με το Ηνωμένο Βασίλειο. Λυπούμε που υπερεύει τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Θαυμάσια τα είπατε, θαυμάσια. Φανταστική ομιλία και ε, πάρα πολύ ακριβείς απαντήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις απαντήσεις που δώσατε και για την ε, διάθεσή σας, την προθυμία σας για συνεργασία. Και εμείς είμαστε διαθέσιμοι και πρόθυμοι και για πολύ σκληρή δουλειά και όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, you see, Ο πρόεδρος Μπούζεκ, πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Όλα βεβαίω πολύ σημαντικά. Και αγαπητές ε, φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εάν επιθυμείτε να μας εγκαταλείψετε που δεν το βρίσκω και πολύ ευγενές, Ω στάση, σα παρακαλώ κάντε το σύντομα. Λυπούμε που το λέω. Θα θέλαμε να αρχίσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αγαπητές φίλε και αγαπητοί φίλοι, το επόμενο θέμα τώρα είναι το υπαρθμόν 7 στην ημερήσια διάταξή μα και προβλέπει την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μαρία Γαβριέλ, Επίτροπο Αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία. Βεβαίω πάντοτε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τα προσφάτως εγκριθέντα νομοθετικά προγράμματα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Χρόνο πολύ δεν έχουμε και βεβαίως το ψηφιακό πρόγραμμα και το ψηφιακό μέρος της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Άρα, ψηφιακό μέρος της διευκόλυνσης και το ψηφιακό πρόγραμμα συνολικότερα. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για μας βεβαίως Μπορούμε να ανοίξουμε συζητήσει και για άλλα θέματα βέβαια, αλλά σας επαναλαμβάνω έχουμε λίγο χρόνο. Γι' αυτό σας παρακαλώ αγαπητές φίλε να είστε σύντομες και θα παρακαλέσω την κυρία Επίτροπο να αρχίσει αμέσως με την εναρκτήρια τοποθέτησή τη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ. σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να προβώ σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας που δείχνει πόση σημασία έχει η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως με την Επιτροπή σας. Θα αρχίσω λέγοντας ότι η καιρή είναι σημαντική διότι αναλαμβάνουμε ε, αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την επόμενη δεκαετία της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σε χρόνο σχετικά περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά οι προτάσεις αυτές οδηγούν σε σημαντικές αναγκαίες αλλαγές για την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό που καθορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός αυτού η ψηφιακή οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο που σημαίνει επίσης σημαντική πρικοδότησή της, χρηματοδότησή της. Με τέσσερα στατικά σημεία για να ανταποκριθεί στις ανάγκες επενδύσεων στον τομέα αυτό. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν όλες τις χώρες μέλη, όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μόνο μέσω μιας κοινή προσέγγισης θα μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ε, ε, ισχυρή και πιο ανταγωνιστική. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την στήριξη του Κοινοβουλίου και εδώ έρχεται η έκκληση για υποστήριξη που σας απευθύνω. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας το όραμα για το μέλλον, τι πρέπει να ζητήσει και να απαιτήσει η Ευρώπη για την ψηφιακή μετάλλαξή της. Πρόκειται για προσπάθεια πολύ σημαντική που ε, ε, εκτελήσεται μέσα στα πλαίσια της Βρετανικής αποχώρησης. Χωρίς τις επενδύσεις κλειδιά, η Ευρώπη και οι συμπολίτε μας θα χάσουμε πολλά πράγματα. Πρώτα, μιλούμε για στήριξη στην ψηφιακή οικονομία. Στήριξη στο ψηφιακό τμήμα μέσα στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στρέφεται γύρω από τέσσερα βασικά στοιχεία. Πρώτα, το νέο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακής καινοτομίας δηλαδή, που εξήγησε προηγουμένως ο κ. Μοέδας, άκουσα ότι ήταν πολύ πλούσια συζήτηση, ο ψηφιακός πυλώνας του μηχανισμού διασύνδεσης της Ευρώπης και τέλος τα μίδια στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Και πρώτα το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη. Τονίζω ότι για πρώτη φορά σε προϋπολογισμό της Ένωσης προτείνουμε πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύσει την αριστεία και την ε, πρωτοπορία της Ένωσης στα ψηφιακά. Θέτοντας αυτά στην ε, υπηρεσία μια ενισχυμένη ανταγωνιστικότητας που θα ωφελήσει όλους. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα είναι διπλασιασμός των όσων πράττουμε υπέρ τη έρευνας και τη καινοτομία. Δεν θα επικαλύπτονται δηλαδή με αυτές τις επενδύσεις. Ο λόγος ύπαρξης του προγράμματος είναι απλός. Πρόκειται για, την, για να διατεθεί στην Ευρώπη η αναγκαία ε, ικανότητα ώστε να μπορέσει να ε, προχωρήσει την ψηφιοποίηση, ώστε η ψηφιακή μεταλλαγή να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτου. Χρειάζεται ταχεία δράση. Γιατί να προέλθει όμως η χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η απάντηση είναι απλή. Η διαπίστωση είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσουν από μόνες τους τις αναγκαίες επενδύσεις. Και για να ακολουθήσουν τέτοιε επενδύσεις σε μεγάλου τομεί της οικονομίας δεν μπορούσε να παραμείνει αυτή η κατάσταση. Επομένως, θα παρεμβαίνει ο, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό για να καλύπτει τα κενά αυτά στι αγορέ για να, αυξήσει το ύψο των επενδύσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι οι ανταγωνιστέ χώρες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποφασίσει να επενδύσουν μαζικά Επομένως, οι χώρες μέλη από μόνες τους δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μαζικές αυτές επενδύσεις στο παγκόσμιο επίπεδο. Μην λησμονούμε ότι ο προϋπολογισμός προτείνει 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στα πλαίσια του τρέχοντος ΠΔΠ, ωστόσο, ιστερεί του προϋπολογισμού των ανταγωνιστών μας. Οποιαδήποτε μείωση θα συνεπάγεται κινδύνους σοβαρούς το ποσό αυτό λοιπόν αποτελεί ποσόν αφετηρίας των επενδύσεών μας. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας για να εκμεταλλευτούμε ε, την ε, ενίσχυση αυτή, να μεγιστοποιήσουμε τις ε, συνεπειές, τις επιπτώσεις της δηλαδή και να διατεθούν οι, οι στηρίξεις αυτές για τις επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες. Το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη θα ενισχύσει τη στρατηγική ικανότητα της Ευρώπης σε τεχνολογικούς τομείς κλειδιά και θα διευρύνει την διάχυσή τους στις, και στο ειδικό τομέα. Θα είναι σημαντική η στήριξη αυτή για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και για να υπάρξει ηγετική θέση της Ευρώπης σε πέντε τομείς. Στην calculating performance, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κυβερνοασφάλεια, στις ε, προηγμένες ψηφιακές ικανότητες και τέλος στην καλύτερη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και την διαλειτουργικότητα. Έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα εν προκειμένου. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από μόνη της θα πρέπει να οδηγήσει σε αυξήσεις πάρα πολύ σημαντικέ του παγκόσμιου ΑΕΠ και εμείς ως Ευρωπαίοι θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο που μας αρμόζει σε αυτό. Το ίδιο σε ό,τι αφορά θέματα κυβερνοασφάλειας, όπου η Ευρώπη πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο και μέσα στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τέλος, σημαντικότερο, η ψηφιακή Ευρώπη, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις ψηφιακές ικανότητε για ευρύτερη χρήση. Για να γίνει αυτό, δείχνουμε την ε, βούλησή μας να κάνουμε την Ευρώπη πατρίδα των ψηφιακών επιχειρήσεων. Λίγα λόγια για το δεύτερο στοιχείο τώρα. Δεύτερο στοιχείο τη χρηματοδοτική στήριξη των ψηφιακών είναι το νέο πρόγραμμα Horizon Europe, Horizon Ευρώπη, του οποίου τα κονδύλια θα αυξηθούν για να φτάσουν τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αναγκαίο μήνυμα για τους ερευνητές και επενδυτές για να συνεχίσουν να χτίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοπορία σε θέματα έρευνας στα ψηφιακά. Θα δώσουμε ξεκάθαρη υποστήριξη στην έρευνα και στην καινοτομία των ψηφιακών τεχνολογιών για να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον τομέα των ψηφιακών και της βιομηχανίας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε γενικές τεχνολογίες όπως για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη ή την ρομποτική στον τομέα της ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας, επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα, στα πλαίσια της ανοιχτή επιστήμης με την υποστήριξη των, τεχνο, ε, ηλεκτρονικών υποδομών και για την καινοτομία, για να ενισχύσουμε τις ε, επαναστατικές καινοτομίες. Αυτά είναι κάποια από τους στόχους που έχουμε θέσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διασύνδεση, ο μηχανισμός Διασύνδεση, δηλαδή το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό ΣΕΦ, χρειάζεται την τεχνολογική υποστήριξη. Με νέο λοιπόν κώδικα για την ηλεκτρονική διασύνδεση και ευχαριστώ πάλι τον πρόεδρο Μπούσεκ και το, τους συζητητές του, κοινο, του Κοινοβουλίου, το μήνυμα που δίνουμε είναι ότι θα διαθέσουμε τα μέσα για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ιδία Σύνδεσης και σε ευχαριστώ πραγματικά για την ε, θαυμάσια συνεργασία. Πάντως ως τώρα, οι επενδύσει δεν ήταν επαρκείς. Δεν αρκούν για να φτάσουμε τους στόχους μας μέχρι το 2025. Θα χρειαζόμασταν 155 εκατομμύρια περισσότερα ευρώ, δηλαδή μέχρι το 2025 για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εδώ πρέπει όλοι να παίξουν τον ρόλο τους και ιδίω στους τομείς εκείνους που έχουν διαμεθοριακή διάσταση και εκεί όπου οι αγορές δεν μπορούν να καλύψουν τα πάντα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας. ΣΕΦ 2, δηλαδή ε, διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, 2 ηλεκτρονική ή ψηφιακή για την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών. Η ψηφιακή μετάλλαξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ο εξυγχρονισμό τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η δημόσια υγεία, όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μια γενικευμένη πρόσβαση σε δίκτυα ε, υψηλής τεχνολογίας. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία υψηλής χωρητικότητας, χρειάζονται νέοι μηχανισμοί που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στις υποδομές της ε, ψηφιακής διασυνδε... διασυνδεσιμότητας. Έχουμε προβλέψει εκεί προϋπολογισμό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το νέο ΣΕΦ θα έχει κυρίως διαμεθοριακή ε, διάσταση. Θα έχουμε δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ε, διαδρόμους πέμπτης γενεάς και προγράμματα τα οποία να οδηγήσουν σε περισσότερη διαθέσιμα gigabyte για τις ε, επικοινωνίες μέχρι και τα σχολεία. Το ψηφιακό ΣΕΦ θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκά δίκτυα πολύ υψηλής δυναμικότητας με, μαζί με το πρόγραμμα ε, Invest EU που θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια υψηλότερη ε, σε μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ε, ψηφιακού κατακαιρματισμού. Το άλλο είναι ο κλάδος των media της Δημιουργικής Ευρώπης, που έχει ως στόχο ιδίω να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού μας τομέα, που εδώ χρειάζεται να επεκταθεί σε περισσότερους τομείς με τεχνολογίες εχμής και η υπεροχή του οπτικοακουστικού τομέα είναι σημαντική πρόκληση και για να ενισχυθούν οι τέχνες αλλά και υπέρ των Ευρωπαίων και για την προβολή των θεμελιωδών αξιών μας των ιδρυτικών θεμελιωδών αξιών μας και εντός της Ένωσης και προς τις τρίτες χώρες. Άρα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν τα θεμέλια της νέας αυτής προσέγγισης για τις επενδύσεις στον ψηφιακό χώρο μέχρι το 2028 για να είναι στέρεες και να αποδώσουν καρπούς σε μια περίοδο όπου θα πρέπει να στηρίξουμε τους σχετικούς προϋπολογισμούς και αναμένω και πάλι και ζητώ την υποστήριξή σας για να δώσουμε στην Ευρώπη την θέση που της αξίζει στην καινοτομία για να ωφεληθεί ολόκληρη Ευρωπαϊκή, όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αναμένω τα σχόλιά σας, τα οποία θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία μου, πάρα πολύ ξεκαθαρά τόσα μα είπατε στην παρουσίασή σα. Δυστυχώ δεν έχουμε τόσο χρόνο και για τα δύο προγράμματα για το Digital Europe και για το SEF, Connecting Europe Facility. Είμαστε βέβαια και για τα δύο αρμόδιοι και βέβαια ιδίω για το θέμα του ψηφιακού πυλώνα του SEF. Και τώρα έχουμε την ε, Αγγέλη Καμπλίνων που είναι η συγγήτρια για το πρόγραμμα Digital Europe, ψηφιακή Ευρώπη. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς, ε, κυρία Επίτροπε, που ήρθατε σήμερα. Είμαι η συγήτρια για το πρόγραμμα αυτό και θέλω να χαιρετήσω την προστάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ θετική. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν ως δέσμευση και ε, έχει, έχει σταματήσει αυτή η ορμή ε, προς την πρόοδο που είχαμε τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το πνεύμα ε, συνεργασίας που επέδειξαν οι υπηρεσίε της Επιτροπής που έπεσε η πρόταση και ήταν, ε, ελπίζουμε ότι και στο μέλλον, στους επόμενε εβδομάδες, μήνες θα συνεργαστούμε με τρόπο αρμονικό. 9,2 δις είναι η σε τρία χρόνια θα ξεκινήσει, υπάρχει πίεση έχουν γίνει ε, πάρα πολλές ε, επαφές και σε τεχνοκρατικό, τεχνικό ε, επίπεδο, οπότε θα πρέπει να τα καταφέρουμε και με αυτή την πρωτοβουλία θα προχωρήσουμε κατά την Αυστριακή Προεδρία, γιατί η Προεδρία αυτή έταξε τα ψηφιακά στις προτεραιότητες του εξαμήνου της. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο όσον αφορά την δυνατότητα να ξεκινήσει μια τέτοια διαδρομή τέλη Ιουνίου, οπότε και εμείς ελπίζουμε να υπάρχει συνεργασία με το Συμβούλιο και όλα να γίνουν όπως πρέπει. Όπως ε, ήδη τόνισε ο Πρόεδρος, είμαστε νομοθέτες και ακριβώς γι' αυτό είμαστε ταγμένοι σε αυτόν τον σκοπό και θα πρέπει να προσφέρουμε στους επενδυτές ένα προβλέψιμο σενάριο για το ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια στην υποστήριξη για όλους τους εμπλεκόμενου και τους εργαζομένους. Οπότε, χάρη στην Επιτροπή, ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά ερωτήματα που εκκρεμούσαν, όμως ακόμη εκκρεμούν κάποια ζητήματα και δεν έπεσαν όλε οι προτάσει ταυτόχρονα, οπότε και παραμένει μια πρόκληση να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με τη συνέργεια μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων, τι θα γίνει με την άμεση διαχείριση των κοινοτικών υπηρεσιών. Οπότε θα πρέπει να σας πω δύο λόγια για αυτό. Πρώτα-πρώτα, super computing. Θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμό και το 2017 είχαμε ε, τις 10 κορυφαίες εγκαταστάσεις super computer, καμία όμως εδώ ε, επίσης ε, ξεχωρίζουν για τέτοιες εγκαταστάσεις ε, δέκα ε, μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εννιά ε, είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο θα αποχωρήσει. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει κάποια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, κάτι το οποίο να προηγηθεί του Τώρα για τη συνέργεια μεταξύ των πυλώνων, για τον συντονισμό μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών. Μπορούμε να προσδοκούμε μια συμφωνία όσον αφορά αυτή την κοινή προσπάθεια. Θα γίνει κάτι τέτοιο σύντομα. Να η πρώτη μου ερώτηση όσον αφορά το super computing τώρα. για την κυβερνοασφάλεια είναι άλλος στόχο, μα είπαν ότι θα υπάρξει ε, μια καινούργια υπηρεσία που θα το αναλάβει. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά πότε θα υποβληθεί η καινούργια σας ε, πρόταση, ποιος δεν είναι ο αρμόδιος ή ενίσα τι αρμοδιότητα θα έχει, πώς θα εμπλέκεται για αυτή τη νέα υπηρεσία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη αυτό απετέλεσε σημαντικό στοιχείο των προηγούμενων πραγμάτων και στη Βαλτική και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι κάνει ο ιδιωτικός τομέας, η συνέργεια ιδιωτικού δημοσίου και σε σχέση με αυτά τα 100 κορυφαία ιδρύματα στην Ευρώπη ε, παραέχουμε πολλές ε, εκθέσεις που λένε ότι είναι έτοιμοι για τις επιχειρήσεις για την νοημοσύνη. Το θέλουν μεγάλες εταιρείες και σχέση με την ιδιοκτησία. Αλλά όχι πλήρως. Να δούμε ποια είναι τα θετικά. Ποιες εφαρμογέ έχουν δοκιμαστεί. Ε, τι γίνεται με τι μικρότερε εταιρείε. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποια hubs, κάποιους κόμβους ψηφιακούς που να καλύψουν τις ΜΜΕ και να βρεθούν τελικά οι λύσει. Όσον αφορά την ανακοίνωση του Απριλίου και το επιπλέον 1,5 δις που επενδύθηκε ε, σύμφωνα με το Horizon 2020 συνεργάστηκε η Κομισιόν τα κράτη-μέλη υπήρξε ένα συντονισμένο πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε τώρα νέους κόμβους για την τεχνητή νοημοσύνη και όταν το 2021 θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, τι θα γίνουν οι υπάρχοντες κόμβοι, θα αναλάβουν νέες λειτουργίες, θα επεκταθεί και σε άλλους στόχους η αρμοδιότητα. Ιδίως όσον αφορά τον οριζόντιο στόχο για τα πιο προχωρημένα, προωθημένα, ψηφιακά ταλέντα δεξιότητες. Και με αυτό το πρόγραμμα τι θα κάνουμε, θα αποτελέσει έναν καταλήτη σε ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο ώστε να έχουμε απορρόφηση της χρηματοδότησης, γιατί ο ρόλος, πάντως, σκοπός δεν είναι να υποκατασταθεί η εθνική προσπάθεια. Δεν θέλουμε να μείνει έξω από το παιχνίδι ιδιωτική επένδυση. Θέλουμε συμμετοχή κάποιων φορέων και από τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα περιορισμό. Αλλά αυτό λέγεται μόνο για το τρίτο στόχο, μόνο για την κυβερνοασφάλεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τι συνέπειε αυτέ, αλλά θα πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την Ένωση όσον αφορά την ευθύνη των τρίτων χωρών που θα συμμετάσχουν στη φάση, στην, στον άξονα τέλο πάντων των κυβερνο, της κυβερνοασφάλειας και τι θα γίνει και με του υπόλοιπου του προγράμματο. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για την πρότασή τη και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία και εγώ και σκιώδη εισηγητέ. Σα ευχαριστούμε για τα όσα μα είπατε για τώρα. η εκπρόσωπη των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ, να... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Επιτροπό. Πρόκειται για ένα κρίσιμο φάκελο για το μέλλον. Αν τα καταφέρουμε η, ψηφιακή είναι η αγορά να γίνει πραγματικά ψηφική, ψηφιακή θα έχουμε κερδίσει. Δεν θα είναι εύκολο. Οι δυνάμεις της αγοράς έχουν αποτύχει σε πολλά σημεία. Δεν θα είναι εύκολο λοιπόν και στην πολιτική εξακολουθούν ή μάλλον οι πολιτικοί εξακολουθούν να επιτρέπουν την δράση πολλών ολιγοπολίων σε πολλές χώρες μέλη. Έχουμε δει ότι οι τηλεπικοινωνίες έχουν κάνει και σημαντικές προσπάθειες ε, στο Wi-Fi. Αυτό βεβαίως οφείλεται και στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ε, telecom, δηλαδή των διαφορών εταιριών τηλεπικοινωνιών. η ΣΤΟΑ, εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει προωθήσει μια στρατηγική που για την ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να γίνει η προσπάθεια μέσα σε σιλό. Το πραγματικός κόσμος αντανακλάται στον ψηφιακό κόσμο. Για μένα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ταυτότητα στον ψηφιακό κόσμο. Για την ώρα γίνεται με μια κάρτα SIM και μια ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση. Αρκούν αυτά για το μέλλον. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε για τη δημιουργία πλατφορμών που θα μας επιτρέψουν, όπως και στην πραγματικότητα, στην καθημερινή πραγματική ζωή δηλαδή, και ε, στην, ε, στον ψηφιακό κόσμο να διασφαλίζεται η ταυτότητα του υποκειμένου κάτι που είναι σημαντικό εκτός από τις δραστηριότητες σάιλο, σιλό και οι pipe activities, δηλαδή οι δραστηριότητες 5G ε, ε, κλπ. πρέπει να επιταχυνθούν και ιδίω ο σχεδιασμός διαμεθοριακών δομών. Η ερώτησή μου είναι, ποια θα είναι η συνεργασία μεταξύ Μπέρεκ, Ενίσα και όλων των άλλων οργανισμών Έχει γίνει κάποια ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ των οργανισμών μας. Έχουμε αρχίσει, ας πούμε, για το machine learning να δούμε ποιοι εργάζονται και ποιοι συνεργάζονται. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει ανάγκη οι οργανισμοί μας να δραστηριοποιηθούν και να συνεργαστούν, γιατί αυτό η σημαντική πρόκληση είναι αυτή η επικοινωνία στην Ευρώπη. Communication Europe. Ο κύριος Σορίνιο. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Είναι σκιώδης εισηγητής. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Αυτό το ψηφιακό πρόγραμμα και λόγω του όγκου πόρων που θα κινητοποιήσει δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μείνει ουραγός ε, να μην υστερεί σε σχέση με μια εξέλιξη που λαμβάνει η χώρα παγκοσμίω. Και εγώ, ως και συζητητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το πρόγραμμα αυτό, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ώστε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρουν να δώσουν συγκεκριμένε απαντήσει και λύσει για του πολίτε. Δεν πρόκειται σε λίγα λεπτά να συζητήσουμε το τόσο πλούσιο αυτό το πρόγραμμα. Θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το ζήτημα τη εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για τόσο δαψιλή ποσά αλλά θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών με την οποία θα συνεργαστούμε να έχει εμπιστοσύνη σε μας. Και ε, θα πρέπει να ζητήσουμε το Wi-Fi for Europe. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσετε το παρόν στην Ολομέλεια του Ιουλίου και να μας κάνετε τη δήλωση για την πρωτοβουλία αυτή. Ε, αλλά ακριβώς είχε μεγάλη απήχηση η πρωτοβουλία αυτή και μας ε, φέρνει ενώπιον των ευθυνών μας. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις δεν μπορούμε στο άρθρο 8 να βρούμε μία λύση για να συνεχίσουμε το Wi-Fi for you ε, ή το Wi-Fi for you too. Θα μπορούσαμε με τα 120 εκατομμύρια που έχουμε για την πρωτοβουλία αυτή να ανταποκριθούμε στο αίτημα των Δήμων, γιατί έχουμε τεράστια ζήτηση από τους ε, Δήμους και για τις υπόλοιπες οντότητες να αφήσουμε το δεύτερο πρόγραμμα, στο οποίο θα αξιοποιήσουμε την ε, εμπειρία που αποκομίσαμε από το πρώτο πρόγραμμα. Νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό ε, κάτι τέτοιο για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί όσο περισσότερη εμπιστοσύνη θα έχουν οι πολίτε στην Ευρώπη, τόσο θα πιάνει τόπο το κάθε ευρώ που θα επενδύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τοσενόφσκι, εκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο Γκαμπριέλ στην Επιτροπή Έρευνας. χαίρομαι που το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε είναι συμβατό με τη δική μου άποψη για τη δομή που θα πρέπει να έχει το ψηφιακό θεματολόγιο. Από την εμπειρία που είχα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ως εισηγητής για το μηχανισμό συνδέοντος της Ευρώπης είναι πόσο εκτενή συζήτηση είχαμε για το ευρυζωνικό διαδίκτυο. Και όσο προχωρούσε ο χρόνος, τόσο περιοριζόταν η φιλοδοξία μας, γιατί δεν είχαμε μια σαφή κατεύθυνση στην πορεία μας. Και συζητήσαμε αυτό το θέμα του διαδικτύου υψηλή ταχύτητα για έξι μήνες εντατικά και μετά από τέσσερα χρόνια το αποτέλεσμα ακόμη δεν είναι σαφές. Σίγουρα η ευρυζωνικότητα είναι μείζον επίτευγμα της Ευρώπης και χρήζει μεγάλης υποστήριξης, αμέριστης όπως μας είπατε κι εσείς. Αλλά θα πρέπει η κατεύθυνσή του να είναι σαφώς προσδιορισμένη. Επίσης, Είμαι σκιώδης ηγετής για το θέμα των υπερυπολογιστών. Και διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα πρόσκομα εδώ. Και η Τσεχία έχει έναν από τους 100 σημαντικότερους παγκοσμίως υπερυπολογιστές. θα πρέπει να δούμε ποιους θα προσκαλέσουμε στη συμμετοχή, για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δαπανούμε μερικές φορές σωστά τα δημόσια κονδύλια με τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο. Επίσης ο χρόνος τρέχει και θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Έχω μία ερώτηση ως προς το σχόλιο σας για το ότι έχει ήδη εξορθολογιστεί η νομοθετική προσέγγιση για, τα, για την ψηφιακή Ευρώπη και έχει ανοίξει ο δρόμος θεσμικά και νομοθετικά. Χωρίς όμως μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις δεν πρόκειται να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Εσείς τι όθηση χρειάζεται ότι θα πρέπει να δώσουμε. Γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά ένα Big bank. Ε, για να πραγματοποιήσουμε ε, πρόοδο στο πρόγραμμα αυτό. Και σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστούμε κύριε Τουσενόφης και ο κύριος Λαλούντα και μέρο των Πρασίνων. Ευχαριστώ. ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπέ. Φαίνεται ότι η πρότασή σας για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη ε, είναι μια αξιόλογη πρόταση και ένα σημαντικό οδικό χάρτη. Έχω κάποιε ερωτήσει. Βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερυπολογιστικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά οι δεξιότητες και οι υποδομές βρίσκονται σε ως δεύτερη προτεραιότητα. Πώς θα αξιοποιήσουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη αν υπάρχουν κενά στο χάρτη ε, διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη και αν υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα και δημιουργεί στρέβλωση και κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς. Η κατάλληλη υποστήριξη για την ανάπτυξη ε, δικτύων ευρυζωνικότητα υψηλή ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλήρη διασυνδεσιμότητα και να ε, γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε, δάσκουμε τα παιδιά μα ε, να ανοίγουν υπολογιστή, να γράφουν έγγραφο ή να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Μπορούμε, τα εκπαιδεύουμε όμω, ώστε να μπορούν να συλλέγουν τι σωστέ ε, πληροφορίε και να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θεωρείται ότι το πρόβλημα αυτό το πραγματεύεστε δεόντως στην πρότασή σας. Επίσης, ε, έχετε την πρόταση της πράξης, ε, ε, της νομοθετικής πράξης για την κυβερνοασφάλεια. Αλλά δεν έχετε τα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης, ό,τι αφορά την πιστοποίηση για την κυβερνοασφάλεια, μερικές φορές γίνεται παραβίαση δικτύου και χρησιμοποιούνται συσκευές εις βάρος των πολιτών. Δεν ε, θέλουμε μια κοινωνία που θα είναι ευάλωτη στο, στην δικτυοπαραβίαση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Κάπελ, εκ μέρους του ΙΕΝΕΦ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς κυρία Επίτροπε. Είστε η πρώτη ψηφιακή επίτροπος που έχει δική της γραμμή. Σημαντικό ε, σύμβολο αυτό για να δείξετε πόσο σημαντικό είναι ο τομέας της ψηφιοποίησης Έχετε βέβαια 9 δισεκατομμύρια μόνο και τα 78% των ε, κονδυλίων αυτών θα πάνε κυρίως σε σούπερ κομπιούτερ, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια. Οι συνάδελφοί μου τοποθετήθηκαν ήδη για τα θέματα αυτά. Βεβαίως ε, χρειάζεστε και την για τι ιδιωτικέ επενδύσει. Για σούπερ κομπιούτερ γνωρίζετε τι γίνεται στην Ασία, γνωρίζετε και τι γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ω τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σωστά ταχθεί υπέρ τη κβαντική τεχνολογία. Και αυτά σχετίζονται πολύ με τα super computer και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει τώρα νέο πολύ ενδιαφέρον δίκτυο. Και στον τομέα τη κυβερνοασφάλεια, ο συναδελφό μου είπε ορισμένα πράγματα ήδη, και θεωρώ ότι ο προπολογισμό του ΕΝΗΣΑ δεν θα είναι επαρκή για να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα τα οποία είναι και αναγκαία και προβλέπονται κιόλα για την κυβερνοασφάλεια. Θα σα παρακαλέσω να δώσετε περισσότερε εξηγήσει και για το τι θα κάνετε και μετά. Ε, ε, εθνικά κέντρα ικανοτήτων. Ίσως μπορείτε να εξηγήσετε σχετικά. Εκτός από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, ακούστηκε σήμερα και το δεύτερο σε σημασία πρόγραμμα στον χώρο της ψηφιοποίησης, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια υπέρ της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη για την διεύρυνση των υποδομών πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι χωρίς την ψηφιακή υποδομή δεν θα καταστεί δυνατόν να γίνουν τα υπόλοιπα βήματα, είτε πρόκειται για την 5G, είτε πρόκειται για το Wi-Fi για όλους τους Ευρωπαίους, η υποδομή για, τα, για τον super computer, όλα αυτά δεν θα μπορέσουν να δημιουργηθούν. Η ΣΕΦ έχει αυξηθεί ο προπολογισμό της κατά 57% και ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί. Ρωτώ λοιπόν, θα λάβετε μέτρα, θα κάνετε βήματα, διότι χρειαζόμαστε ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων για την δημιουργία ε, έργων υποδομής διαμεθοριακών. Θα έρθετε σε επαφή με τις χώρες μέλη για να καταδείξετε την αναγκαιότητα μιας ε, διεύρυνσης των ε, δικτύων που θα μεταφέρουν τα σήματα 5G. Το επίσημο, πρόγραμμα που μας αφορά για τον επόμενο προϋπολογισμό ε, ε από περισσότερους πόρους. Ε, το ξέρουμε, πρόκειται για μια επίσημη πρόταση η οποία εγκρίθηκε στην Επιτροπή μας. Α, επομένως είναι σημαντικό αυτό να ληφθεί υπόψη, συνάδελφοι. Όλοι οι υπόλοιποι. Άλλοι δύο έχουν εγγραφεί. Ο Ντουάρ Μαρντέν και ο Γιώργο Μιρόβλητσεκ. Μάρτεν, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε και εσάς κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση. Πάρα πολύ γρήγορα καθησυχάστηκε 100% γιατί ε, ε, ε, ακόμα και όσον αφορά τα ψηφιακά που είναι της αρμοδιότητας μας όπως είπατε νομίζω ότι πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα και ότι αυτό το κείμενο για την κυβέρνηση ασφάλεια για το φιλτράρισμα των επενδύσεων είναι πέρα από αυτά τα οποία πρέπει εμείς να απαιτούμε οπότε η κυβέρνηση αφορά όλες τις χώρες αλλά δεν ξέρω εάν μπορούν οι χώρες να έχουν τα μέσα που χρειάζονται για να έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Οπότε ακόμα και αν είναι πέρα από εμάς το να παρέμβουμε στον προπολογισμό, ε, να μην το προσφέρουμε αυτό, έχοντας υπόψη για το τι γίνεται με την ε, Κίνα, γιατί κοιτάνε προς τα εδώ, προς την Ευρώπη, να δουν μπορούν να αγοράσουν κάποιες εταιρείε, ιδίως όσον αφορά τα ψηφιακά ε, υψηλή δεξιότητα, ε, εξειδίκευση κλπ. Οπότε έτσι θα πρέπει αυτό να το έχουν υπόψη και τελευταίο να σας ρωτήσω για αυτό το bug του, για το wifi fi στην Ευρώπη, γιατί μπλοκαρίστηκε. Είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε στην επόμενη τον Οκτώβριο. Ε, ήταν λίγο τεχνική αντιμετώπιση. Όποιος προλάβει και είπαμε ότι υπήρχε κάποιο είδους λαθροχειρία τι θα γίνει, θα συνεχίσετε στην ίδια βάση ή θα το κάνετε πιο επαγγελματικά στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς συνάδελφοι. Α, ο κύριος Κόχλης, μία και μόνο ερώτηση. Πώς θα έχουμε ταχύτητα ταχύτητας σε όλη την Ευρώπη, για το έχουμε όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε. Μόνο αυτά από πλευρά μα Αναμένονται οι απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν τον λόγο. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τόσα ρωτήθηκαν. Πρώτα-πρώτα, με τη σειρά ενωπημένη σε γκρουπ Ναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Λίναρ, το ότι θα συνεργαστούμε. Είχαμε δήματα ε, διευκρίνησης και ερωτήσεις και για τα δύο προγράμματα είχαμε ερωτήσεις, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε με 7 κρατημέλη, τώρα έχουμε 20. Και θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Και με την Βουλγαρική Προεδρία θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το joint undertaking, γι' αυτό και εγώ σας το λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για την διακυβέρνηση, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή, όλα αυτά δεν τα ξεχάσαμε και είναι σημαντικό για μας να μην αφήσουμε στην άκρη της ΜΜΕ και δεν θα πρέπει να είναι θέμα μιας ελίτ, θα πρέπει να είναι θέμα ε, λίγων. Θα πρέπει να ωφεληθούν όλες οι ΜΜΕ και με το πρόγραμμα θα έχουμε 2,7 δις ευρώ Ούτως ώστε να αποκτήσει άργα και οστά αυτή η πρωτοβουλία μέχρι το 2023. Έχουμε στατευτεί γι' αυτό, θα ε, κάνουμε επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιους κανόνες θα ρυθμιστεί αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα για τους Digital Innovation Hubs, χρηματοδοτούμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν μέσω του κόμβου και στο μέλλον για το Digital Europe θα έχουμε το πρώτο πρόγραμμα για τη δημιουργία αυτού ή αυτών των κόμβων. Οπότε σε κάθε μέλος να υπάρχει ένας λειτουργικός κόμβος και να δούμε στη συνέχεια πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δούμε τι θα κάνουμε αυτούς τους κόμβους και να έχουμε μέχρι το 2020 παντού τέτοιους κόμβους. Υπάρχει ένα αυθεντικό δίκτυο μεταξύ αυτών των κόμβων και έτσι μην έχουμε επικαλύψεις, μην έχουμε επαναλήψεις. Να μπορέσουν επίσης να ρίξουν το βάρος της Ε. Πριν γίνει η απόφαση για την επένδυση να έχει γίνει δοκιμή. Α, κάτι που είπε η κυρία Λίναρ. Τι γίνεται με τις ε, ψηφιακές δεξιότητες, πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θεωρήσουμε ότι θέλουμε έναν κόμβο σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης, ξέρουμε ότι για να υπάρξουν οι δεξιότητες έχει μεγάλη σημασία το θέμα της εγκύτητας για τους Ευρωπαίους. Οπότε αυτό μας απασχολεί, με και το επιτολίο μου και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική και θετική η συμβολή του Κοινοβουλίου για την κυβερνοασφάλεια τώρα. Καταρχήν, ο ρόλο του Οργανισμού Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Είναι σαφώ προσδιορισμένο. και μην ξεχνάμε ότι ο ΕΝΙΣΑ υπάρχει και έχουμε την, την οδηγία ΕΝΙΣ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ήδη από το Μάιο. Θα δούμε πώ θα εφαρμοστεί, γιατί αυτή η οδηγία είναι η πρώτη νομοθετική πράξη που έχουμε για την κυβερνοασφάλεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΙΣΑ, τον Οργανισμό Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, υπάρχει και λειτουργεί. Θέλουμε να ενισχύσουμε πάντως τις ικανότητε του ΕΝΙΣΑ και τις ε, λειτουργικές, τις επιχειρησιακές, αλλά και τον προπολογισμό του ΕΝΙΣΑ. Και όταν μιλώ για επιχειρησιακές ικανότητε. θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι στην πρότασή μα προβλέψαμε τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να ζητήσουν από τον ΕΝΗΣΑ να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τα τροτά σημεία τους και να δουν πώς θα τα διορθώσουν. Οπότε σίγουρα ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ δεν θα έχει ρόλο πέραν της εντολής που διαθέτει. Σε ό,τι αφορά τη μία ενό νέου οργανισμού, όχι δεν μιλούμε για νέο οργανισμό, για νέα αντότητα, μιλούμε για τη δημιουργία ενός κέντρου ε, δεξιοτήτων ή αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη με ένα κεντρικό συντονιστικό φορέα, ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οπότε στην πρόταση για τον ΕΝΙΣΑ προβλέπεται ένα τμήμα του προσωπικού του οργανισμού ε, να εδρεύει στις Βρυξέλλες για επιχειρησιακούς σκοπούς, ώστε να εξασφαλίζει αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ του ΕΝΙΣΑ και των υπόλοιπων οργανισμών. Τώρα ξεκινά αυτή η συνεργασία ήταν ε, ε, σαφώς κάτι που δεν το είχαμε αναφέρει μέχρι τώρα. Και μέσα σε ένα μήνα και κάτι ήδη υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του σεφ ε, του Europol, του ΕΡΕΝΗΣΑ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ακριβώς για να προβλέψουμε δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη αντοχή μας και αθεκτικότητά μας για την κυβερνοασφάλεια. Μίλησα με τον Διευθυντή του ΕΝΙΣΑ και είναι κάτι που το ε, επισημαίνω επανειλημμένος όταν συζητούμε μαζί. Ακριβώς επειδή υπάρχουν νέες τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτός ο συντονισμός και η συνεργασία το συντομότερο δυνατόν. Και το θέμα αυτό θα με απασχολεί μονίμως. Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη και το πρόγραμμα Wi-Fi for You, γιατί είναι αλληλένδετα τα δύο σημεία. Τι συνέβη καταρχήν με το πρόγραμμα Wi-Fi for You. For you. Όντως, ε, το ομολογώ ότι γίναμε τα θύματα της επιτυχίας μας. Ουδέποτε δεν είχαμε τόσο ζωηρό ενδιαφέρον από τους Δήμους για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τέτοια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου ήμασταν τα θύματα της επιτυχίας μας. Σε λιγότερο από ένα μήνα είχαμε 18.000 εγγραφές και στις 15 Μαΐου όταν έγιναν τα επίσημα εγγένεια λάβαμε 3.500 εγγραφές τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα τα 10 δευτερόλεπτα, τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα 5.000 εγγραφές και τότε ένα τρίτο μέρος μας ενημέρωσε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και μερικοί μπόρεσαν να, ε, να υποβάλουν υποψηφιότητα πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε αναγνωριστεί. Γιατί όταν είναι μία στις Βρυξέλλες, στη Βουλγαρία είναι δύο η ώρα. Και σε αυτό δεν φταίνε οι Δήμοι. Αλλά χωρίς να το ξέρουν, κατάφεραν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους πριν τα επίσημα εγγένεια. Άλλοι μετά. Και η αρχή μας είναι, προλάβει, είναι η σειρά προτεραιότητα, όποιο προλάβει. Και δυστυχώ δεν συνέτρεξαν οι προποθέσει για να τηρηθεί αυτή η αρχή της σειράς προτεραιότητας, το οποίο προλάβει. Οπότε, ε, κρίναμε σκόπιμο να ακυρώσουμε αυτή την πρώτη ε, έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά ε, μεριμνήσαμε ώστε να μην μείνουμε πίσω, να μην έχουμε καθυστέρηση. Γιατί αν είχαμε συνεχίσει την έκκληση για την υποβολή ενδιαφέροντο όπω έγινε στι 15 Μαου, οι χίλιοι πρώτοι υποψήφοι θα έπρεπε να λάβουν την ε, κοινοποίηση το Σεπτέμβριο. Τώρα αυτό το πρόγραμμα κρατούμε. Θέλουμε το φθινόπωρο να έχουμε και πάλι το διαγωνισμό και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Δήμους που ήδη έχουν εγγραφεί ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους, γιατί ήδη είναι εγγεγραμμένοι. Απλώς θα ζητήσουμε να πατήσουν το κουμπί submit, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους και προσπαθούμε με το επιτελείο μου να αποφύγουμε επανάληψη αυτού του προβλήματος και ακριβώς επειδή συνέβη μια φορά κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο και είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε περισσότερα μέσα για να καλύψουμε περισσότερους δήμους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σίγουρα να είστε βέβαιοι για την υποστήριξή μου, ώστε να έχουμε και Wi-Fi 2. Αλλά πρώτα να ε, λειτουργήσει το πρώτο, το πρώτο πρόγραμμα, γιατί σας ε, ομολογώ ότι στεναχωρήθηκε, γιατί πραγματικά είχε συμβολικό χαρακτήρα αυτό το σχέδιο. Πάντως, το Σεπτέμβριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερους δήμους που θα λάβουν το κουπόνι και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουμε ε, να υποστηρίζουμε ένα σχέδιο που ε, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το προωθήσω όσο μπορώ. Και έχω εμπλακεί και προσωπικά στο θέμα αυτό Λυπάμαι για αυτό που συνέβη, πάντως ε, δεν χάνουμε τον ενθουσιασμό μας ότι τη θέση μας θα φροντίσουμε να μην επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, ένα θέμα που όπως ξέρετε μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Στο πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη προβλέψαμε 500 εκατομμύρια ευρώ για τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Και γνωρίζετε τα νούμερα καλύτερα από μένα. Αυτή τη στιγμή μας ε, λείπουν 350.000 ε, ειδικοί, ε, στο μέλλον θα μας λείπουν 500.000 εμπειρογνώμονες και σίγουρα ε, αυτό το κενό δεν το καλύψουμε μόνο με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Γι' αυτό θέλουμε συντονισμό και με άλλους επιτρόπους, για παράδειγμα με το πρόγραμμα Erasmus Plus, με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή παιδεία και μέχρι τον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε το πειραματικό σχέδιο για τις ψηφιακές δυνατότητες και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε 5-6 φοιτητές στην Ευρώπη να κάνουν διασυνοριακά στα μαθητείας 4 με 5 μήνες και έχουμε ήδη 450, 450 προσφορές από επιχειρήσεις 350 με 500 προσφορές από επιχειρήσεις και θέλω και εσείς να φροντίσετε στις χώρες σας να γίνει γνωστή αυτή η πρωτοβουλία για να προσελκύσουμε φοιτητέ που δεν είναι μόνο ε, φοιτητέ ε, σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνίας, αλλά και σε κοινωνικές επιστήμες, σε επιστήμες ε, της ζωής, για να ασχοληθούν με την υπερυπολογιστική, το blockchain, το web design και σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή παιδεία, ήδη εκεί προβλέψαμε το Wi-Fi for you για τα σχολεία και δημιουργήσαμε κάποια προγράμματα και για τους διδασκάλους, για το διδακτικό προσωπικό. Γιατί σήμερα πάνω από 25% των νέων λένε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους καθηγητές τους γιατί δεν γνωρίζουν καλά τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό το κενό θα πρέπει να το καλύψουμε, αυτή την πρόκληση να την αντιμετωπίσουμε ε, σε συνδυασμό και συνεργασία με άλλους επιτρόπους, να ενισχυθούν οι δεξιότητες και των καθηγητών. Και σίγουρα δεν ε, ε, έχουμε κάνει ιεράρχηση μεταξύ της τεχνικής νοημοσύνης ε, και των δεξιοτήτων ή της δημόσιας διοίκησης και της υπερυπολογιστικής. Πέντε είναι οι τομείς ε, στους οποίους θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο ταυτόχρονα και γι' αυτό προτείνουμε τις σχετικές στρατηγικές επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υποδομές και τις ταχύτερες διαδικασίες, προς το παρόν δεν μπορώ να δεσμευτώ, αλλά το έχουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις, τις λευτικές ζώνες ε, ή τα κενά, τη διαφορά μεταξύ αστικών και κέντρο και υπαίθρου. Ε, έχουμε το θέμα του ΣΕΒ, έχουμε τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού από ένα στα τρία δις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το νέο κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών γιατί για να έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις θέλουμε νομική προβλεψιμότητα, ασφάλεια των επενδύσεων και γι' αυτό ακριβώς ε, επενδύουμε στον κώδικα, νέο κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με μέτρα συνδυασμένων επενδύσεων ώστε να διαμορφώσουμε ένα καλό πλαίσιο για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη ισορροπία που θα μπορούσαμε να βρούμε μεταξύ των τριών οργάνων για το αρχικό κείμενο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, την τεχνητή νοημοσύνη, και ένα κέριο ζήτημα φυσικά, θα ήθελα να πω ότι στη στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε εντοπίσει τρεις ισότιμες διαστάσεις κατά τη γνώμη μας. Καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε τις βιομηχανικές και τεχνολογικές ικανότητες και γι' αυτό χρειαζόμαστε επενδύσεις. Ο στόχος είναι σαφής. 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι το 2020. Επίσης, ε, κινητοποιώντας ταυτόχρονα δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια, θα μπορούσαμε μέχρι το 2020 να έχουμε 20 δις και στόχος είναι να έχουμε 20 δισεκατομμύρια το χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Δεύτερο σημαντικό σημείο στη στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας και το θέμα των δεξιοτήτων. Και γι' αυτό η κόμβη ψηφιακής καινοτομία και το blueprint, το μηχανισμός ώστε να αντιμετωπίσουμε την ε, τομεακή ζήτηση πολύ πιο γρήγορα είναι σημαντικά θέματα. Και τρίτη πτυχή της στρατηγικής μας για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτή είναι και προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, είναι το θέμα το ηθικό, διοντολογικό και νομικό. Και εκεί έχετε προχωρήσει, γιατί η κυρία Ντελβό έχει ήδη συντάξει την έκθεσή της και έχουμε ε, συστήσει μια ε, ομάδα υψηλού επίπεδου με 52 εμπειρογνώμονες και για πρώτη φορά έχουμε ομάδα εργασίας και με εκπροσώπους των κρατών μελών και Είχα προηγουμένω συζήτηση μαζί του πριν έρθω στη δική σα επιτροπή και είναι σαφέ για όλου ότι όταν μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται για μοναδική ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονό ότι οι πολίτε φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά του και δεν έχουν ακόμα εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αυτά τα θέματα των δεξιοτήτων, των κόμβων ψηφιακή καινοτομία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης έχουμε μια πλατφόρμα για την καταπαραγγελία τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε μια τέτοια πλατφόρμα για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και πρόσβαση σε αλγόριθμους. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία λοιπόν. Πάντως για την τεχνητή νοημοσύνη ε, υπάρχει μια σημαντική όθηση και μαζί με τα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη συμφωνούμε ότι πραγματικά θα είναι ευκαιρία για την Ευρώπη να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία της και την ηγετική της θέση. Αλλά θα πρέπει να οριοθετήσουμε ε, την δική μας προσέγγιση χωρίς να αδιαφορούμε για τα ηθικά, διοντολογικά, κοινωνικο-οικονομικά θέματα και τα ζητήματα των δεξιοτήτων. Και σίγουρα θα συνεργαστούμε με την κυρία Λίναρτ, την εισηγητριά σας, για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν κατάφερα να εξαντλήσω όλες τις ερωτήσεις. Ελπίζω να μην παρέλειψα τίποτα. Το τελευταίο θέμα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας και πάλι και το θέμα της πιστοποίησης. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, ολοκληρώνει το δικό του έργο αυτή τη στιγμή για το θέμα της πιστοποίησης. Εμείς είχαμε προτείνει προαιρετική, εθελοντική βάση. Και όταν μιλούμε για κυβερνοασφάλεια, δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα στα χέρια των κρατών μελών, στη δική τους διακριτική ευχέρεια. Γι' αυτό και έχουμε συγκεκριμένο ρόλο του οργανισμού ΕΝΙΣΑ. Έχουμε το σύστημα πιστοποίηση που προτείνουμε για πρώτη φορά και όπου οι βιομηχανίε και τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν. Και επίση, όταν μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια ω δυνατότητα, ικανότητα ανθεκτικότητα σε επίπεδο κρατών μελών, Περιμένω να δω πώς τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν τη στρατηγική, το blueprint, το μηχανισμό συντονισμού για, μεγάλη, για μεγάλες κλίμακες επιθέσεις και πώς θα γίνει επιχειρησιακή αυτή η στρατηγική. Εγώ περιμένω να έχουμε κέντρα αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη με ένα κέντρο αριστείας στις Βρυξέλλες για να επενδύσουμε στην εμπειρογνωμοσύνη και να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές ώστε να ενισχύσουμε την πρόληψη και την αθεκτικότητά μας και να μην καλούμαστε εκ των υστέρων να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Αυτά και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θαυμάσια τα είπατε. Και δεν έχουμε βέβαια πολύ χρόνο. Δώσατε όμως ακριβείς απαντήσεις και σας ευχαριστώ αναμένουμε συνεργασία μαζί σας στο μέλλον. Έχουμε πράγματι πολύ δουλειά μπροστά μας. Αύριο, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 10 προβλέπονται ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας. Θα σας δω αύριο και καλό σας βράδυ.